Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ που είσαστε ακριβείς και είσαστε εδώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιες σύντομες ανακοινώσεις του Προέδρου. Πιστεύω ότι ξέρετε κάποια πράγματα, διότι το είχα προανακοινώσει χθες. Ανταλλαγή απόψεων με το στατηγό Μοριγιών προβλεπόταν για σήμερα το απόγευμα ακυρώθηκε λόγω απεργίας τρένων εις Γαλλία και Βέλγιο και ανεβλήθη λοιπόν αυτή η συνάντηση για τη συνέδριαση της 10ης Νοεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα και θα είναι τότε εκτός του κύριο Μοριγιών και ο κύριος Μπερμάν, συνάδελφος Μπερμάν που διορίστηκε επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών για τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών που ακυρώθηκαν διότι απεσύρθη ο αντίπαλος του Καρσάη, ο Αμπτουλά Αμπτουλά. Γι' αυτό ήθελα να μην θυσιάσουμε εντελώς την ε, συνεδρίαση το το σήμερα και να βάλουμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή το 13 που αφορά τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες ε, μετά από τις πρωινές εργασίες. θα κλείσουμε τις εργασίες μας με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στο τέλος των εργασιών των πρωινών θεμάτων. Μετά που η Τσεχία επικύρωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας, αφού έγινε αυτό και έχει επικυρωθεί ουσιαστικά η συνθήκη της Λισαβόνας και ο διορισμός των επιτρόπων, του το εκπροσώπου και των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι κάτι που να γίνει στο τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα, πρέ, θα εμπλακεί άμεσα ή έμεσα στην διοργάνωση κάποιων ε, ακροάσεων, επιτρόπων, της διεύρυνσης, ανάπτυξης, ε, διεθνούς εμπορίου και βέβαια πρώτα απ' όλα ε, και θα ασχοληθεί και με το θέμα των αντιπρόεδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του είπα το εκπροσώπου που ο ύπατος εκπρόσωπος ήταν ουσιαστικά υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τις εργασίες Επιτροπής μας. Αν δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις όσον αφορά το καθορισμό των χαρτοφυλακίων των Επιτρόπων, αυτές οι ακροάσεις θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Στρασβούργου για την ε, θέση του, της ανάπτυξης και του Διεθνούς Εμπορίου του Επιτρόπου για αυτά τα θέματα. Και την επόμενη εβδομάδα, αρχές Δεκεμβρίου, θα γίνει μια κανονική τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη, ε, για τη συνέχεια των διεργασιών αυτών. Οι ημερομηνίε θα σας ανακοινωθούν το ταχύτερο δυνατόν, οπότε είναι δυνατόν. Όμως θα πρέπει να σημειώσετε ήδη την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο ημερολόγιο σας που προβλέπεται για την ακρόαση του ΙΠΑ του εκπροσώπου και των αντιπρόεδρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει προβλέψει η διάσκεψη των πρόεδρων. Έχει υπάρξει συμφωνία όσον αφορά αυτή τη ημερομηνία. Λοιπόν, παρακαλώ, σημειώστε τι. Μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη πρόταση ψηφίσματο. Ορίστε. Κύριε Άτκινς, συνάδελφε Άτκινς, διαδικαστικό, συγγνώμη, όσον αφορά τι διευθετήσει αυτέ τι διοικητικέ. Θα εκτιμάτε βεβαίω ότι είναι πολύ αργά τώρα να μας λέτε ότι θα γίνει μια κρόαση Παρασκευή. Είναι πολύ άβολο αυτό, πάρα πολύ άβολο για συναδέλφους που έχουν δεσμεύσει στι εκλογικές τους ε, ε περιφέρειες και άλλε αντιμέ υποχρεώσει. Βλέπω ότι γνέφεται και εσεί έχετε δύο πρόβλημα. έχω μια δέσμευση και δεν πάω ξεφύγω εύκολα εκείνη την ημέρα, διότι κανονικά δεν συνεδριάζουμε την Παρασκευή. Δεν υπάρχει παραμικρή δυνατότητα να αλλάξει αυτή η ημερομηνία. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούμε δυστυχώς. Έχετε δίκιο και εγώ έγνεφα διότι ήθελα να πω αυτό, να εκφράσω αυτή τη σκέψη, τη μοιράζομαι και εγώ όπως όλοι μας τις πρώτες και τελευταίες ημέρες της εβδομάδας έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, στην εκλογική μου περιφέρεια. Εναλλακτική ποια είναι ότι δεν θα καταφέρουμε να δούμε τον είπατε πρόσωπο και τον αντιπρόεδρο πριν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτή την επιλογή του μεταξύ διαβόλων διαλέξαμε και διαλέξαμε το διαβολάκι αν θέλετε. Και είναι μια απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, οπότε μπορώ, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Βλέπω τον κύριο Χάουιτ και με τον κύριο Πόσελτ που θέλω το λόγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με τη σειρά. Πρώτα είδα τον κύριο Χάουιτ, μετά εσείς, κύριε Πόσολτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να είναι θέμα με κατανόησης. Είπατε ότι ο εκπρόσωπο είναι είναι μπορεί να είναι Ο, ε, ο, μπορεί να είναι ο ή και γυναίκα. Εγώ υποστηρίζω τον David Miliband. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χ, το ο, το αρσενικό, εντάξει, υπό τι πρώτε περιστάσει στη γενική έκφραση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρσενικό άρθρο. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει. Υπάρχουν και κάποιες εκδοχές λεξιλογίου που σε κάποιους ρόλους ε, δίνουν στο φίλο στα Ιταλικά. Είναι μόνο θηλυκό. Και η τίγρη είναι μόνο θηλυκή στα Ιταλικά. Παρόλο που υπάρχει και ο τίγρης. Καμιά φορά επικρατεί ένα φύλλο στο λεξιλόγιο. Τέλο πάντων. Λαμβάνω υπόψη αυτά που είπατε. Ο κύριο Πόσολτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βάζουμε διάφορα πράγματα και ε, την Παρασκευή. Καταλαβαίνω βέβαια και τη θέση των συναδέλφων που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις και ιδίω πρώτων Χριστουγέννων. Έχουμε πρώτη Δευτέρα και τρίτη Δεκεμβρίου τριήμερη, τριήμερο συνεδριάσεων. Και θέλω να μάθω εάν αντί για τη συνεδρίαση δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ακρόαση. Γιατί και να μην είναι δυνατόν. Και εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο αποφάσισε έτσι η ε, διάσκεψη των Προέδρων. Καμιά φορά νομίζω ότι δεν αποφασίζουμε σωστά κριτήρια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν από εκείνους που καθόρισαν την ημερήσια διάταξη και δυνατότητα να επιλεγούν μέρες οι πιο βολικές για όλους εξετάστηκαν. Υπάρχουν ακροάσεις άλλων επιτρόπων που δεν επικαλύπτονται, δεν επικαλύπτουν τι άλλε υποχρεώσει μα και έχουν ελεύθερη, αφήνουν ελεύθερη την Παρασκευή και λυπάμαι. Αλλά εδώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση, εναλλακτικέ, πιο πρακτικέ και βολικέ δεν βρέθηκαν. Δεν βρήκαμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την σε διάταξη. Πρόταση ψηφίσματο σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009. Η συγητής είναι ο κύριος Βόμποντα που επισκέφθηκε τις δύο χώρες, τη Σλοβενία και την Κροατία πρόσφατα και του δίνουμε το λόγο για να κάνει παρουσίαση στο θέμα. Ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να έλθω σε λίγα συγκεκριμένα θέματα. Χθε έγινε ήδη μια συζήτηση που περιέλαβε πολλά θέματα. Ένα από αυτά που συζητούνται ξανά και ξανά είναι το θέμα του συστήματος δικαίου και του αγώνα κατά της διαφθοράς. Στον τομέα αυτό έχει επιτύχει σημαντικές πρόοδους η Κροατία. Πάντως δεν έχει καλύψει όλο το δρόμο που θα έπρεπε. Τονίζω και στην έκθεσή μου ότι αυτά τα θέματα ειδικά πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και να ενισχυθεί η προσπάθεια που κάνει η κροατική κυβέρνηση. Τελευταία παρετήθηκε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ήρθε η ασυλία του προηγούμενου Υπουργού Αμήνης. Εγώ δεν θα προβώ σε καμία κρίση για τα πρόσωπα αυτά, γιατί δεν μου αρμόζει κιόλα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρξαν παρετήσει, παρέτηση δηλαδή, και άρση τη ασυλίας, αποτελεί ένα μήνυμα και για μένα, αλλά και για του ε, Κροάτες πολίτες, ότι κανεί δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι πρόσωπα τα οποία επί των οποίων επικρέμαται κάποια υποψία πρέπει εν τέλει να αχθούν και ενώπιον των δικαστηρίων. Δεύτερο. Διαπιστώσαμε ότι η θετική απήχηση στα λαϊκά στρώματα υπέρ της ένταξης δεν είναι τόσο υψηλή όσο θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε. Συζητήσαμε χθε ότι και διάφορες κοινωνικές ομάδες, ακόμη και η Εκκλησία, επέκριναν, επέκριναν αυστηρά τις συμφωνίες με την Σλοβενία και ότι θεωρούν ότι η ένταξη ή θα πρέπει να γίνει μετά από κάποια συνένεση με τη Σλοβενία ή καλύτερα να μην γίνει καθόλου. Εν πάση περιπτώσει εδώ χρειάζεται να γίνει πολλή ενημέρωση και διαφώτιση. Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με το ποινικό δικαστήριο της Χάγης και αυτό το θίξαμε χθε. η κροατική κυβέρνηση έχει ιδρύσει μια ομάδα ειδικών καθηκόντων, μια special task force και προσεκάλεσε και τον Βάιμερτς να συμμετάσχει με εκπροσώπους του στην ομάδα αυτή αλλά και εκπροσώπους άλλων χωρών μελών ως παρατηρητές για να δουν εάν και κατά πόσον η Κροατία αναζητεί τα έγγραφα εκείνα τα οποία ακόμη αξιώνει να δει το δικαστήριο. Ο εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου δεν θέλει να αναμειχθεί, αλλά υπάρχουν χώρε μέλη οι οποίε μπορούν να στείλουν εκπροσώπου σε αυτή την ομάδα ειδικών καθηκόντων για να παρακολουθήσουν, να παρατηρήσουν και να διαπιστώσουν εάν πράγματι εργάζεται με τον καλύτερο τρόπο η ομάδα αυτή. Την πρόσκληση την έκανε η ίδια η κροατική κυβέρνηση και νομίζω πρέπει να την δεχθούμε. Δεν γίνεται κατανοητό από πλευρά Κροατία ότι αφενό υπάρχουν κριτικέ που λένε ότι εσεί οι Κροάτε κάνετε πολύ λίγα πράγματα. Από την άλλη μεριά, όταν βγαίνουν οι Κροάτε και λένε Ελάτε, στείλτε μα ειδικού να παρακολουθήσουν τι εργασίε που κάνουμε, τότε δεν ανταποκρινόμαστε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ να ανταποκριθούμε. Τώρα, επιστροφή προσφύγων κλπ. Βεβαίω εδώ υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα και ιδίω σχετικά με εκείνου του εσωτερικά εκτοπισμένου οι οποίοι επιστρέφουν, οι οποίοι ίσω δεν είχαν κάποια περιουσία, αλλά ίσως είχαν κάποιο, ε, κάποια κοινωνική στέγη η οποία τους αφαιρέθηκε και τώρα αναγκάζονται να ζήσουν χωρίς καμία αποζημίωση. Προσπαθεί να δώσει κάποιες λύσεις η Κροατία, γίνονται κάποια βήματα, κάνει δηλαδή προσπάθεια να ε, δώσει λύσεις. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τον ανταγωνισμό, ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το θέμα των ναυπηγείων, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό, ότι πρέπει να γίνει δεύτερη διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν νομίζω το θέμα αυτό πρέπει να παρεμποδίσει την ένταξη. Πρέπει ωστόσο να υλοποιηθούν ορισμένα πράγματα και εκεί. Τώρα για τις δημόσιες προμήθειε. Ακόμα δεν είμαστε πεπισμένοι ότι τα πράγματα πηγαίνουν εκεί όπως θα έπρεπε. Βέβαια και σε ορισμένε χώρε μέλη διαπιστώνονται παρασπονδίε. Πάντω η Κροατία πρέπει να φροντίσει ώστε οι διαδικασίε αυτέ να είναι διαφανεί, ανοιχτέ και να υπακούν σε ξεκάθαρου κανόνε. Για το τέλο, τελευταίο θέμα είναι η περιφερειακή συνεργασία και οι διμερείς σχέσει. Ήδη χθε συζητήσαμε το θέμα της συμφωνίας με τη Σλοβενία. Οι δύο πρωθυπουργοί την υπέγρασαν επιτέλους εχθές. Μένει ανοιχτό το θέμα της κύρωσης της συμφωνίας αυτής. Εγώ έχω περιλάβει και μία επιφύλαξη, ε, τέλο πάντων μία παρατήρηση. Η λίστα που πρόκειται να συντάξει η Κομισιόν σχετικά με τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο δικαστήριο αυτό θα πρέπει να είναι ε, προσωπικότητες με ιδιαίτερα προσόντα οι οποίες να έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Και παρακαλώ να δεχτείτε το κείμενο όπως είναι στην πρώτη έκδοση της ε, συμφωνίας όπου λέει δηλαδή να γίνει ένας επίσημος κατάλογος που θα συνταχθεί από τον πρόεδρο της Κομισιόν. Θα διαβιβάσω το μεταφρασμένο κείμενο στους συναδέλφους. Το άλλο καλό είναι ότι η Κροατία ανέλαβε την πρωτοβουλία να <coughs> επιλύσει διαφορές με άλλους γείτονες που δεν ήταν τόσο βαρύνουσες, με τη Βοσνία Ζιγοβίνη δηλαδή, για παράδειγμα, την οποία προσεκάλεσε μέσα σε διμερείς συμφωνίες, διμερεί ε, συνομιλίες να, γίνει, ε, να δοθεί κάποια λύση. Με το Μαυροβούνιο έχει πάει τώρα στο ε, Διεθνές Δικαστήριο τη Χάγης. Πρόκειται για μια σημαντική για μας διαπεριφερειακή συνεργασία για μια επίλυση διμερών προβλημάτων που πρέπει μέχρι τέλους των διαπραγματεύσεων να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να είναι δυνατόν, κατά τη γνώμη μου, οι διαπραγματεύσει να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Εάν βέβαια αποδώσουν πράγματι οι προσπάθειες της κρατικής κυβέρνησης και αν επιληθούν τα ε, προβλήματα που μένουν ακόμη ανοιχτά. Δεν είναι δικό μας καθήκον ε, να κρίνουμε εν προκειμένου αλλά νομίζω θα χρειαστεί και μια ε, περίοδος κυρώσεως Τη συμφωνίας, της, ε, συμφωνίας ένταξης που θα κρατήσει ένα-ένα μισή χρόνο. Πάντως, όπως είπα, θεωρώ ότι μέσα στο 2010 μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό θα καταστεί δυνατόν, όπως είπα, εάν είναι επιτυχής οι προσπάθειες που καταβάλει η κρατική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Μόνο μία διευκρίνηση εφόσον αναφερθήκατε στο κείμενο που διανεμήθη. Είναι μια προσωρινή εκδοχή διότι αυτή που ελέγχεται από τους, νομομαθ, τους γλωσσομαθείς νομομαθίστα είναι έτοιμοι μαζί με τη μετάφραση, όταν μεταφραστεί το κείμενο. Δηλαδή, αφορά η παρατήρησή σας και αυτό που προβλέπονται να γίνουν. Ο κύριος Πόσελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον κύριο Σβόμποντα για την πραγματικά για άλλη μια φορά διαβιέστατη αλλά και σύντομη έκθεσή του και επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι ευρωβουλευτές εδώ θα ήθελα να τους απευθύνω έκκληση σε όλους δηλαδή τους συναδέλφους μακάρι όλοι και όλες να διατηρήσουμε αυτό το στυλ των εκθέσεων και να είναι το κείμενο λιτό και σύντομο και να μην χώνουμε μέσα παν το επιστητό. Διότι έχουμε και την έκθεση πλαίσιο του πρόεδρου μας Αλμπερτίνη που αναφέρεται στη στρατηγική. Τότε λοιπόν α μην μπαίνουν μέσα πράγματα τα οποία ισχύουν ούτως ή άλλως και για πολλές χώρες μέλη και για ε, πολλούς, πολλές υποψήφιες χώρες. μην μπαίνουν λοιπόν τα πράγματα αυτά μέσα. Α περιορίζονται οι εκθέσει, η περιοριστεί παρούσα έκθεση στην εξέταση τη πραγματική παρούσα κατάσταση της Κροατίας. Αυτό το πράττει η έκθεση με θαυμάσιο τρόπο και νομίζω ότι πράγματι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει το 2010, χωρίς βεβαίω να είναι δεσμευτικός ο στόχος αυτό Μπορούμε να το βάλουμε στην έκθεση ωστόσο, για να μην έχει την εντύπωση και η Κροατία ότι προσπαθούμε να ε, κάνουμε κάποιες καθυστερήσεις. Σωστά είπε ο κ. Φόποντα ότι αρχίζει και υπάρχει κάποια επιφύλαξη μέσα στον κρατικό πληθυσμό απέναντι στην ε, ένταξη. Δεν αρκούν οι προσπάθειες της κρατικής κυβέρνησης για να ξεπεραστεί η επιφύλαξη αυτή. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποια προσπάθεια. Διότι έχει την εντύπωση ο κόσμος εκεί ότι καθυστερεί και καθυστερεί, αναβάλλεται και αναβάλλεται. Ότι βεβαίως πρέπει να πληρωθούν τα κριτήρια είναι σαφές. Στο ΖΙΤΑ ε, στο G έχει ένα continuous. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θέμα το οποίο ε, επιτρέπει κριτικές ότι δηλαδή έχουν την εντύπωση οι Κροάτες ότι πάμε να εφαρμόσουμε άλλα κριτήρια από ό,τι σε άλλες υποψήφιες χώρες. Για παράδειγμα, η επιστροφή των προσφύγων. Πήγα στην Βοηβοδίνα, δηλαδή στη γειτονική περιοχή της ε, Σερβίας και ρώτησα έναν δήμαρχο «Έχετε στην πόλη σας ακόμα Κροάτες πρόσφυγες» και μου απάντησε ότι όλοι έχουν επιστρέψει πλέον. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα, αλλά σε σύγκριση με την κατάσταση σε άλλε γειτονικέ χώρε υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επιστροφή προσφύγων στην Κροατία και σε άλλε χώρε. Κάτι τέτοιο πρέπει να το αναγνωρίσουμε και πρέπει να εκφράσουμε την αναγνώριση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο τη Χάγη. Πάλι εδώ πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουν. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένε χώρε μέλη πάνε τώρα να διορθώσουν κάποια σφάλματα που έχουν κάνει στο παρελθόν και αυτό αποβαίνει σε βάρος της Κροατίας. Όταν άρχισε ο πόλεμος τότε το 99 όλοι ξεκίνησαν, όλοι έκαναν λάθη. Τώρα πάνε κάπως να τα διορθώσουν με τρόπο υπερβολικό. Και αυτό συζητείται στην κοινή γνώμη της Κροατίας και θα έπρεπε να είμαστε δίκαιοι να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της Κροατίας. Κανείς δεν μιλάει πλέον για τον στρατηγό Μλάντιτς. Τον έχουν όλοι σχεδόν ξεχάσει. Όμως παρακολουθούν όλοι με το μεγεθυντικό φακό τις προσπάθειες που κάνει η Κροατία και τις κρίνουν ή τις επικρίνουν. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορώ να σας συστήσω να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα με τρόπο ευαίσθητο. Το πράττει αυτό ο κύριος Όποντα. Και να ζητήσουμε ώστε μέχρι τέλους του έτους το αργότερο αρχέ του επόμενου έτου να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια και οι δυνατόν να κλείσουν το πολύ μέχρι τα μισά του επόμενου χρόνου. Ευχαριστώ λοιπόν τώρα και πάλι τον κύριο Σβόμποντα. Βρίσκω την έκθεσή του εξαιρετικά ισορροπημένη. Έχει κριτικό χαρακτήρα, αλλά πραγματικά έχει και την δυνατότητα να ε, βοηθήσει, να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Σωστά προσαρμοστήκατε στην, ε, αναφερθήκατε στη σαφήνεια του συγητού και στο πόσο σύντομο ήταν και επειδή όλοι ε, πάρα πολύ θέλω να μιλήσουν. Έχουμε 11 αναφερθούμε σε τρεις εκθέσει. γι' αυτό παρακαλώ να παραμείνετε εντός του ορίου των τριών λεπτών τη παρέμβασης. Κύριος Κάτσιν έχει το λόγο. Ελπίζω για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πρώτα συγχαρητήρια στον κύριο Σφόμποντα για το σχέδιο ψηφίσματος. Ο κύριος Σφόμποντα απέδειξε ότι είναι γνώστης του θέματος αλλά είναι και πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα καθήκοντά του. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο κύριος Πόσελτ, αλλά παρόλα αυτά θέλω να επισημάνω τα συμπεράσματα της χθεσινή συζήτηση, ότι δηλαδή παρόλη την υπογραφή τη συμφωνία μεταξύ Σλοβενία και Κροατία ακολουθεί μια κρίσιμη φάση και αυτό διότι χρειάζεται να υπάρξουν οι πλειοψηφίες για την κύρωση της συμφωνίας. Η Κροατία έχει το δικαίωμα να δώσει στον εαυτό της χρόνο ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει αυτή τη συνένεση μεταξύ του κυβερνώντος συνασπισμού και της αντιπολίτευσης. Τώρα, για την παράγραφο ε, G, όπου λέει ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το, τα μέσα του 2010. Ε, ε, Αυτό βρίσκω δεν είναι σωστό. Είναι δύσκολο να τηρηθούν τέτοιες προθεσμίες. Είναι καλύτερα να συμφωνήσουμε να βάλουμε μια γενικότερη διατύπωση, για παράδειγμα, το ταχύτερο δυνατό. Διότι η Κροατία είναι εκείνη η οποία θα κρίνει εν τέλει ε, τι είναι δυνατό και τι όχι. Διότι αν βάλουμε ε, μια ημερομηνία θα θεωρηθεί σαν εξαναγκασμός από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία καταβάλει προσπάθεια, έχει ένα δυναμισμό και θεωρώ ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει. Αλλά είναι καλύτερα να βάλουμε μια γενικότερη διατύπωση παρά μια προθεσμία η οποία ενδεχομένω να μην μπορέσει να τηρηθεί. Πάντω, θα συστήσω στον κύριο Σφόμποντα στην παράγραφο του 27 όπου σωστά τονίζει ε, τα καθήκοντα που πρέπει ακόμα να επιτελέσει η ε, Ιουγκοσλαβία αναφέρεται και στην κληρονομιά της ε, πρώην Αυτή είναι δύσκολη ε, υπόθεση και πολυμερής που όμως και για την Κροατία και για τις γειτονικές χώρες και κυρίως για εκείνες οι οποίες ακόμα δεν έχουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας μέλους. Για όλες αυτές τις χώρες λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ταυτόχρονα επισημαίνω μια ε, απαράδεκτη πρακτική που είναι στη, υπάρχει στην ε, ε Κροατία. Δηλαδή καταδικάζεται κάποιο για εγκλήματα πολέμου και ξαφνικά εξαφανίζεται. Δεν ανεβρίσκεται πλέον στην Κροατία διότι έχει μεταβεί στην Βοσνία και εκεί ε, αισθάνεται ασφαλής. Αυτά πρέπει να λεχθούν. Εξάλλου υπάρχει το ε, κτηματολόγιο το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο και είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κόλλημα για την επιστροφή των περιουσιών των εκτοπισμένων. Ευχαριστώ κύριε Κάτσιν. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπρόκ, συντονιστή του ΕΛΚ, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Συγχαίρω με τη σειρά μου για την έκθεση του κ. Σφόμπαντα και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την υπογραφή της συμφωνίας χθες στην Στοκχόλμη μεταξύ των δύο πλευρών. Και ελπίζω τα όσα μόλις είπε ο κύριος Κατσίν να μην σημαίνουν ότι θα προκύψουν νέες δυσχέρειες. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου διμερεί θέματα, διμερή θέματα να μην παρεμποδίζουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αντίθετα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί την βάση για την επίλυση. Διότι αλλιώ έχουμε ε, το σύνδρομο αυτού που βρίσκεται ήδη μέσα στο λεωφορείο και λέει «Α, εγώ είμαι μέσα, να μην σταματήσει το λεωφορείο για να πάρει κι άλλους». η Κροατία ως μη χώρα μέλος δεν ευρίσκεται στην ίδια θέση να μπορέσει να προβάλλει ενδεχομένως θεμητές απαιτήσει απέναντι σε άλλη χώρα μέλος, διότι, απέναντι σε χώρα μέλος δηλαδή, διότι δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα χώρα μέλος. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται παρακολούθηση. Γι' αυτό θα έρθω και σε αυτό που είπε και ο κύριο Πόσελτ για την συνεργασία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Η έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων με την Κροατία ήδη καθυστέρησε σημαντικά επειδή ε, ε, ανεζητεί το κάποιο ο οποίο δεν ήταν καν πλέον στην Κροατία αλλά βρέθηκε τελικά στα Κανάρια νησιά. Σε αυτό επιμένουν ακόμα ορισμένε χωρισμένοι. Έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι εγκαταλείπεται η αρχή του ότι πρέπει κάθε χώρα να κρίνεται ανάλογα με τα όσα έχει επιτύχει και μπαίνουν συγκρίσεις με άλλες ε, χώρες μέλη, με άλλες μάλλον υποψήφιες χώρες και, και γίνονται διασυνδέσεις με τις συνταξιακές πορείες άλλων χωρών. Αυτά δεν μπορούν να έχουν ωστόσο αποφασιστικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων. Στην έκθεση του κύριο Σφόποντα, λέει ότι υπάρχουν θέματα της δημόσιας διοίκησης, υπάρχουν θέματα διαφθοράς. Μας τα είπε και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Κροατίας χθες στη συζήτηση, ότι δηλαδή χρειάζεται ακόμα να κάνουν σοβαρές προσπάθειες. Και ότι αυτές οι προσπάθειες δεν γίνονται για χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να τα κάνουν ούτως ή άλλως οι Κροάτες, ακόμα και δεν ήθελαν να γίνουν ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ωφελήσουν την ίδια τους τη χώρα. Ο κύριος Βόμποντα μιλεί και για την περιορισμένη απήχηση της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά τα πράγματα αυτά, οι προσπάθειες αυτές της εξυγίανσης πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως. Και όχι, όπως είπα, για χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις ε, χωρών που ήταν υποψήφιες και εντάχθηκαν, πρέπει να επιμείνουμε ώστε οι Κροάτε να επιταχύνουν τι προσπάθειε αυτέ και οι δυνατόν διαπραγματεύσει να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Η κυρία Πάκ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπροκ με κάλυψε. Εγώ απλώ θα κάνω τις διατυπώσεις του ακόμα λίγο πιο αυστηρές. Σε ευχαριστώ, Έλμαρ, που τα είπε. Υπενθυμίζω ότι ιδίω στην δικαιοσύνη μετά από τη νέα κροατική κυβέρνηση πριν από 1,5 χρόνο και με, την, ε, ε, με τον νέο αστυνομικό διευθυντή και ούτω καθεξής επέτυχε σημαντικές πρόοδους. Όντως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντως οι Κροάτες βρίσκονται σε καλό δρόμο. Τονίζω επίσης ότι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αντιμετωπίζεται με τρόπο ανεύθυνο, διότι χρησιμοποιείται το επιχείρημα αυτό με ε, στόχο να καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσει. Δεν θα πω ποια χώρα είναι αυτή, αλλά υπάρχει μια χώρα η οποία επιμένει ξανά και ξανά ότι δεν ε, συνεργάζονται οι Κροάτες πλήρως με το δικαστήριο της Χαγή. Κάθε πρόσωπο που αναζητήθηκε τελικά βρέθηκε, ακόμα και αν βρισκόταν στην Βεντούρα. Τώρα αναζητούνται κάποια έγγραφα. Πρόκειται για, ένα, για έγγραφα που, ε, ε, που βγήκαν από την διεξαγωγή ενός πολέμου. Ήταν ένας αστραπίος πόλεμος, ο οποίος έγινε και ήταν και επιτυχής. Ορισμένα έγγραφα ίσως να μην υπήρξαν καν. Είμαι βέβαια, άλλωστε, ότι ορισμένα καταστράφηκαν εκ των υστέρων. Αυτό το έχει διαπιστώσει και η, κροατική, και η κροατική κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση η οποία τότε δεν ασκούσε τα κυβερνητικά κοθέκοντα και τώρα έρχεται και διαπιστώνει ότι ορισμένα έγγραφα δεν μπορούν να βρεθούν πλέον. Ή ίσω μάλιστα και καταστράφηκαν. Το πολύ που μπορεί να κάνει είναι να τιμωρήσει αυτόν που τα κατέστρεψε. Δεν φταίει όμω η ίδια κυβέρνηση επειδή έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχουν πλέον τα έγγραφα που αναζητεί το δικαστήριο. Τώρα, για το έτο 2010. Δεν λέμε στην έκθεση ότι το 2010 θα πρέπει η Κροατία να γίνει χώρα μέλος. Λέμε ότι μέσα στο 2010 μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Και θα παρακαλέσω τους ε, Σλοβαίνους να μην είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Ας μην ξεχνούν ότι από το 1998 είχαν την προοπτική ότι το 2004 θα γίνονταν μέλος ακόμα και αν δεν είχαν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια. Και έγιναν μέλος το 2004 και η διαδοχή της πρώην Ιουγκοσλαβία να μην ε, ενταχθεί στην έκθεση μόναχα για την Κροατία. Και οι ίδιοι οι Σλοβαίνοι ήταν μέρος της ε, ε, πρώην Ιουγκοσλαβία. και μιλώ για την Λιουμπιάννα Μπάτκα. Μην φορτώνετε όλα σας τα προβλήματα στην γειτονική σας χώρα. Κανένας δεν το έπραξε σε βάρος σας, μην το κάνετε κι εσείς τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πακ. Βάιγκελ, επόμενο αγορητή για τρία λεπτά. Κύριο Βάιγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εκπλήσωμαι. Πώς, πώς εξελίσσεται αυτή η συζήτηση για την Κροατία. Διότι Φιλίες όπου δεν ασκείται καμία κριτική, καμιά φορά βλάπτουν παρά να ωφελούν. Νομίζω ότι η τελευταία παρέμβαση το παράκανε. Ξεφεύγει από τα κοινοβουλευτικά έθιμα. Και παρακαλώ να όταν μιλείτε για τη Σλοβενία να μιλείτε αντικειμενικά και για το θέμα της διαδοχής και σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Σλοβενίας για την ένταξη της Κροατίας. Η Σλοβενία πάντοτε υποστήριξε την Κροατία στην ενταξιακή της πορεία και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Δεν χρειάζεται να μας ενθαρρύνεται εντό εισαγωγικών με τέτοιε παρατηρήσει. παρατηρήσεις. Για τον κύριο Σφόμποντα θα πω ότι θα συμφωνήσω διότι βρίσκω την προσέγγιση του πολύ ισορροπημένη διότι η έκθεσή του περιέχει και επένους αλλά και κριτικές οι οποίες είναι απαραίτητες. Και εγώ θα κάνω ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις οι οποίες έχουν πιο πολύ τον στόχο να δώσουν μια όθηση. Για παράδειγμα, η επιστροφή των Σέρβων στην Κροατία είναι πολύ δραματικότερη από αυτά που ακούμε σήμερα και που ακούσαμε και χθε. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραμείνει από τον πόλεμο και χρειάζεται κάποια ευαισθησία και η Κροατία πρέπει να τα αντιμετωπίσει και αυτή με κάποια περισσότερη προσοχή και περισσότερη ευαισθησία. Το δεύτερο, το είπε ο ίδιο ο κύριος Κατσίν, πρόκειται για το θέμα ότι ένας καταδικασμένος εγκληματίας πολέμου μπορεί, εφού και να έχει ακόμη καταδικαστεί, μπορεί να μεταβεί σε μια γειτονική χώρα, να καταφύγει εκεί και παρόλα αυτά να παραμείνει μέλος του κρατικού κοινοβουλίου. Μιλώ για την περίπτωση Γκάρας. Και το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι το γεγονός ότι η Κροατία εμπλέκεται σε όλες τις εξελίξεις και τις εκλογές στη γειτονική Βοσνία. Και το αντίθετο, όταν εκλέγεται η Κροατική Βουλή. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα και οδηγούν σε αποσταθεροποιήσεις και προβλήματα. Τα οποία μάλιστα τονίζουν και ορισμένα κροατικά κόμματα, τα οποία δεν ωφελούνται από την κατάσταση αυτή. Εν τέλει, θέλω να πω ότι η ανάμιξη της Εκκλησίας στα πολιτικά στην ε, Κροατία και η αυστηρή καταδίκη από πλευρά της Εκκλησίας της συμφωνίας με τη Σλοβενία πρέπει να καταδικαστεί. Ευχαριστώ κύριε Βάγκερ. Λούνατσεκ, το επόμενο όνομα που στο κατάλογο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Κυρία Λούνατσεκ. Υπάρχουν βέβαια τα γνωστά διμερεί προβλήματα μεταξύ Κροατία και Σλοβενίας. Δεν θα επισέλθω σε αυτά. Μέχρι τώρα νομίζω η συζήτηση κινήθηκε με συλλογικά πλαίσια. Θεωρώ την έκθεση του κ. Σόμποντα εξαιρετική και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα. Πρόκειται για ένα ορθό μείγμα μιας κριτικής στάσης, πολύ σωστά, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν προβλήματα τα θέτει και ιδίω στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και άλλα βέβαια, και παρόλα αυτά διαφαίνεται μέσα από την έκθεσή του η υποστήριξη που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ενταξιακή πορεία της Κροατίας. Θα αναφερθώ σε τρία θέματα. Το ένα συζητήθηκε και χθε στη συζήτηση με τον Κροάτη Υπουργό Εξωτερικών και ίσω πρόκειται για αυτή την περίπτωση σκάνδαλο της αντιμετώπιση μιας μη κρατική οργάνωση, της Friends of the Earth οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μπροστά σε ένα κρατικό υπουργείο και όπου η νέα κρατική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την οργάνωση αυτή, Friends of the Earth, με το νέο περιβαλλοντικό δίκαιο, πηγαίνοντα να του επιβάλλει ένα πρόστιμο βαρύτατο 50-100.000 ευρώ, κάτι το οποίο σημαίνει το τέλο τη οργάνωση αυτή. Ο ίδιο Υπουργό Εξωτερικών χθε είπε ότι θα επιληθεί το θέμα του μόλι επιστρέψει στην Κροατία. Εγώ θέλω να προτείνω, εάν δεν ξεκαθαριστεί η υπόθεση και εν πάση περιπτώσει αν δεν μια θετική λύση στο θέμα αυτό στι επόμενε εβδομάδε, να περιλάβουμε μια προσθήκη στην τροπολογία 1 για την παράγραφο 25 που αναφέρεται στο περιβάλλον όπου να λέμε ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εφαρμόζεται το νέο περιβαλλοντικό δίκαιο και ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται το δίκαιο αυτό για να αποτρέπει ή να τιμωρεί ε, διαμαρτυρίες και διαμαρτυρόμενους για θέματα περιβάλλοντος. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ευχάριστο το ότι και ο Χάνες Φόμποντα θέτει τα θέματα ε, που υπάρχουν με ε, τις ε, μειονότητες. Αυτά με τη σερβική μειονότητα, τα προβλήματα που είχαμε με τη σερβική μειονότητα είναι τώρα πλέον λιγότερα. Υπάρχουν όμως και οι Ρώμα. Και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα, είναι η μειονότητα των ομοφιλοφίλων. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί εδώ που θα συμφωνήσουν μαζί μου, αλλά η διάκριση σε βάρος ε, της ε, ε, ερωτικής ας πούμε είναι κάτι το οποίο διαπιστώνεται εντονότατα στην Κροατία. Και εν τέλει, μία φράση κύριε Πρόεδρε ακόμα. Η Κροατία παίζει ένα θετικό ρόλο και στη Βοσνία για τους Κροάτες που διαβιούν εκεί. Και θα ήθελα να περιεχθεί και εδώ μια τροπολογία, να ζητηθεί δηλαδή από την Κροατία να συνεχίσει να παίζει ένα σταθεροποιητικό ρόλο για την ενίσχυση και τη συνταγματική ενίσχυση δηλαδή του κράτους της Βοσνίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ο κ. Σαγκουράκης έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω να κάνω τι εξή παρατηρήσει στην έκθεση που παρουσίασε ο κύριο ε, Σφόμποντα. Ε, καταρχήν θέλω να σα διευκρινίσω ότι μιλάω εξ ονόματο του κόμματό μου και όχι εξ ονόματο τη ομάδα GUE-NGL, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω. νομίζω ότι το κοινοβούλιο μα θα έπρεπε να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι δεν μα πείθει ποια θα είναι τα ωφέλη για τους εργαζόμενους και γενικότερα για το λαό της Κροατίας από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας είναι προφανές ότι θα είναι ελάχιστα, ή θα υπάρχουν καθόλου ωφέλη. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που θα ωφεληθούν θα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεγάλα πολυεθνικά μονοπόλια, που ούτως ή άλλως έχουν μια μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή και βλέπουν και αυτή τη χώρα, όπως πολλές άλλες χώρες της ε, ε, Ανατολικής Ευρώπης ως νέους τομείς δραστηριότητας και αποκόμισης κερδών. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο, όπως σημειώνεται και στο σχέδιο ψηφίσματος, υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση στη χώρα όσον αφορά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντίθεση θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω μιας αντιδημοκρατικής διαδικασίας για την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να προτείνω, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα ο λαός της Κροατίας, αν το θέλει φυσικά, να αποφθανθεί με δημοψήφισμα, τουλάχιστον στο θέμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωμα που δεν είχε να εκφράσει όταν τέθηκε το θέμα ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και μιας και έγινε λόγος για διακρίσεις και ε, κινητοποίηση ενάντια σε ε, ε, αντιπολίτευση, θα ήθελα να ενημερώσω το Ευρωκοινοβούλιο ότι πριν δύο χρόνια γίνανε διαδηλώσει, οι οποίε εκφράζαν την αντίθεση μερίδα του πληθυσμού τη χώρα ένταξη του ΝΑΤΟ και το αποτέλεσμα ήταν περίπου το ίδιο με αυτό που μα περίγραψε η συνάδελφο πριν. Ε, παραπέρα. Συγκεκριμένα στο σχέδιο ψηφίσματο του κυρίου Σφόμποντα θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη στο σημείο ε, εκεί που γίνεται λόγο για τη συμφωνία μεταξύ Κροατία και Σλοβενία, αυτή η συμφωνία να τεθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να ε, επικυρωθεί μόνον και να επικυρωθεί μόνον με ε, απόφαση του ΟΗΕ. Αλλιώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπως η απόσχηση του Κωσόβου με τα προβλήματα που έχουμε. Τέλος, ανησυχώ πάρα πολύ για το σημείο 12 του σχεδιού ψηφίσματος που αν δεν προσθεθεί ότι οι όποιες διαδικασίες δεν πρέπει να οδηγήσουν στην αναθεώρηση των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα ανοίξει μια πολύ επικίνδυνη και άσχημη κατάσταση όχι μόνο στην Κροατία αλλά και γενικότερα. Και τέλος, τα ζητήματα των συνόρων αγαπητοί συνάδελφοι δεν είναι διμερεί ζητήματα. Είναι ζητήματα διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου μόνο στη βάση αυτή μπορούν να λύνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Τρία λεπτά για τον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ τρία λεπτά. Άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά την έκκληση του κυρίου Πόσελτ. Έκκληση προς τους ευρωβουλευτές να είναι σύντομοι στις παρεμβάσεις τους και ακριβείς. Να πω ότι θα έπρεπε ο κύριος Πόσελτ να εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια και στον εαυτό του κυρίως όσον αφορά το κείμενο ψηφίσματος που προτείνει ο κύριος Βόμποντα. Το κείμενο είναι καλά ισορροπημένο και εμπνέει την Κροατία να είναι θαραλέα. Γι' αυτό προτείνω να υιοθετήσουμε το κείμενο όσο έχει. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Μία απάντηση ζήτησε να δώσει ο κύριος Πόσελτ να δευτερολογήσει. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είπα ότι ε, πρέπει να είμαστε ε, σύντομοι γιατί πράγματι κανένας δεν με πιστέψει άμα το πω εγώ. Είπα να μην ε, βάλουμε τροπολογίες γιατί το ίδιο το κείμενο του Κυριού Σβόμποντα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά να πω δύο πράγματα τώρα. Για το πρώτο, κύριε Λούνατσεκ, κυρία Λούνατσεκ, ε, για αυτά μιλούσα για ε, θέματα μη διακρίσεων που νομίζω ότι δεν εντάσσονται εδώ διότι δεν είναι ε, επί της ουσίας, συμφωνώ μαζί σας αλλά δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε κάθε μια από τις εκθέσεις είναι, ε, υπάρχει έκθεση πλαίσιο που είναι για όλες τις ε, υποψήφιες χώρες μπορούν να μπουν τα πράγματα αυτά εκεί γιατί για τα θέματα μη διακρίσεων η Κροατία είναι υποχρεωμένη να δεχτεί το κοινοτικό κεκτημένο, επομένω να εφαρμόσει ό,τι εφαρμόζουν και οι υπόλοιπε χωρισμένοι. Δεύτερο, ε, ο προβληματισμός ή το πρόβλημα Κροατίας-Σλοβενίας. Κύριε Βάγκελ, θυμηθείτε, έγινε ο πόλεμος τότε δεν ε, επετέθη η Κροατία κατά της Σλοβενίας. Ο Ιουγκοσλαβικός στρατός επιτέθηκε καταρχής, κατα, ε, ε, καταρχάς κατά της Σλοβενίας και μετά κατά της Κροατίας. Βρισκόσασταν λοιπόν στο ίδιο, στην ίδια μοίρα τότε και για τη Συμφωνία Συνδέσεως. Είχαμε πει τότε, αν είχαμε πει τότε ότι η Κροατία θα μπορέσει να ενταχθεί μόνο όταν θα επιληθεί το θέμα των συνεργατικών διαφόρων, αν το είχαμε πει τότε αυτό και για την Σλοβενία, δεν θα υπήρχε σήμερα το θέμα. Όπω λοιπόν είπε και κάποιο άλλο συνάδελφο προηγουμένω, α μην είσαστε βασιλικότεροι του βασιλείου. <coughs> Καλώ. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Δύο λεπτά. Κύριο Βάγκελ θα δευτερολογήσει. Δεν χρειάζομαι δύο λεπτά, θα ήθελα ένα λεπτό μόνο. Συνεχίζει στα γερμανικά. Συμφωνώ μαζί σας ότι και η Κροατία και η Σλοβενία υπήρξαν θύματα επίθεσης και στρατιωτικής εισβολής μιας ε, ενός τότε δικτατορικού ε, ε λαϊκού στρατού αλλά η Σλοβενία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχεδόν λιμένα τα συνοριακά προβλήματα με την Κροατία στη βάση της τότε συμφωνίας και το σημείωσε αυτό τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφορά όταν λέω δηλαδή ότι το συνοριακό θέμα είναι σημαντικό για την ένταξη. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Η κυρία Αλεξάνδρα Καστχράνχε. Ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας. Ελπίζω. Είσαστε ένας από τους λίγους που προφέρει σωστά το όνομά μου. Να σας πω ότι είναι η τρίτη μέρα στη δουλειά και η δεύτερη μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για δεύτερη φορά έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, βλέπετε ποιες προτεραιότητες έχω να είμαι εδώ να σας ακούω. Έχω κάποια σχόλια. Από ό,τι βλέπω από τη συζήτηση τη σημερινή, βλέπω ότι εν γέννη είναι κοινό ο στόχος μας. Δηλαδή η, Κροατία να φτάσει στη λήξη των διαπραγματεύσεων σύντομα με καλά αποτελέσματα και να πληρούνται όλα τα κριτήρια. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Και καλά πάνε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω. Η συμφωνία της 10 ε, η Σεπτεμβρίου ήταν πάρα πολύ ε, καλή για να ανοίξουν τα έξι κεφάλαια και να κλείσουν άλλα πέντε. Η χθεσινή υπογραφή είναι ακόμα ένα σημαντικό βήμα. Το θέμα αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για τη Σλοβενία, την Κροατία και την ε, Ένωση αυτή η συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουμε και τι δύο χώρε να προχωρήσουν προ την κύρωση ε, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις. Χθε ήταν η μέρα εορτασμών και πανηγυρισμών, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε προ το μέλλον, να φτάσουμε στο τέλο, να γίνει η κύρωση. Να λήξουν διαπραγματεύσει, πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα η Κροατία σε διάφορου τομεί, αυτό αναφέρεται στην έκθεσή μα. και το αναφέρατε πολλοί από εσά σήμερα. Ποιοι είναι οι βασικοί, όλοι οι τομεί αυτοί είναι στον πολιτικό τομέα. Ε, Δικαστικό τομέα, δημόσια διοίκηση, καταπολέμηση διαφθορά και οργανωμένου εγκλήματο, μειωνοτικά δικαιώματα και επιστροφή των προσφύγων, εγκλήματα πολέμων, δίκες και πρόσβαση στα διάφορα έγγραφα του διεθνούς, για το Διεθνές Δικαστήριο. Τονίζει η έκθεση ότι υπάρχει δέσμευση για την καταπολέμηση της Χρειάζεται αύξηση του δυναμικού της κυβέρνησης για αυτόν τον σκοπό και της διοίκησης. Ας το δούμε και από άλλη πλευρά. Υπάρχει πολιτική δέσμευση και η βούληση, αλλά όχι σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να διαπνέει όλη την κοινωνία, όλη τη διοίκηση και βελτιώθηκε το δυναμικό της διοίκησης. Οι δυνατότητες της διοίκησης βελτιώθηκαν. Γίνονται αλλαγές και περιμένουμε για τα αποτελέσματα. Πολιτική βούληση και δέσμευση υπάρχει. Αλλά πρέπει να ε, περάσει όλα τα επίπεδα. Για το πρόβλημα των προσφύγων να πούμε ότι αυτό είναι που είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι το πρόβλημα των εσωτερικών προσφύγων εντός της χώρας, αλλά των προσφύγων που έρχονται από άλλες χώρες, που πρέπει να έρθουν κάποια στιγμή. Υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα για τη στέγαση αυτών και πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά τις πρόσφυγες. Για το θέμα ICT πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο κυρίως το κεφάλαιο 23. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις και επειδή λείπουν έγγραφα και αν δεν δοθούν στον αρμόδιο φορέα στο δικαστήριο τα έγγραφα, θα ακολουθήσουμε λάθο δρόμο. Πρέπει να γίνουν τώρα πολλά πράγματα σε αυτό τον τομέα. Η Κροατία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να παραδώσει ε, στο δικαστήριο τα έγγραφα. Δεν ξέρω μέσω τη ομάδα Cruises Task Force με άλλο τρόπο δεν ξέρω να φτάσουν τα έγγραφα στο δικαστήριο. Η έκθεση αυτή θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλά ισορροπημένη, καλή διατύπωση, ταιριάζει και με πρώτερες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ευχαριστούμε μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Δεν ξέρω αν η θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ να είσαστε σύντομο. Διότι σίγουρα έχουμε περάσει το χρόνο που είχαμε διαθέσει για αυτή την έκθεση και έχουμε μπει στο, στα χωράφια άλλων εκθέσεων. Μία πληροφορία και μία έκκληση. Η πληροφορία για τον συνάδελφο που απορρίπτει την ένταξη. Στην Κροατία υπάρχει δημοψήφισμα. Εφόσον απορρίπτεται κάτι, τουλάχιστον να είστε ενημερωμένο. Θα έχει λοιπόν ο κροατικό πληθυσμό τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Δεύτερο, για του συναδέλφου. Οι δύο πρωθυπουργοί υπέγραψαν χθε μια συμφωνία. Υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ Κροατία και Σλοβενία και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε πολέμους χαρακομμάτων. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε, να βασιστούμε σε αυτό το καλό κλίμα για να βοηθήσουμε και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν και γρήγορα στην ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Κάποιες πληροφορίε όσον αφορά τα διαδικαστικά προθεσμία υποβολής τροπολογιών 8 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία 26-27 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας και το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους που πήρατε το λόγο. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2009. Η Ζόραν Ζόραν Τάλερ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, όπως είπα και πριν, αν μπορείτε να τηρήσετε τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι και εγώ βρέθηκα στα Σκόπια για δύο ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα και η ε, παρουσία μου εκεί με βοήθησε πολύ για τη σύνταξη της ε, έκθεσης διότι μπόρεσα να γνωρίσω την παρούσα κατάσταση. Μπόρεσα και συναντήθηκα με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο της Βουλής, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και με σημαντικές προσωπικότητες των κομμάτων στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή με όλα τα πρόσωπα εκείνα τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις. Στην... Τα πρόσωπα δηλαδή τα οποία υποτίθεται ότι με τις προσπάθειές τους θα βοηθήσουν την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να προχωρήσει ε, στην πορεία μιας ένταξης κάτι που νομίζω ότι θα ήταν και το καλύτερο για την χώρα αυτή. Έχουν λοιπόν επιτελεστεί σημαντικές πρόοδοι και έχουν ε, υπάρξει και κάποιες οψιοδρομήσεις. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας έχει εκπληρώσει τα κριτήρια για την ε, διευκόλυνση των προξενικών θεωρήσεων. Μέσα Οκτωβρίου ήρθε και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την πλήρη ένταξη. Οι διπλωματικές σχέσεις με το, με το γειτονικό Κόσοβο έχουν ε, ε, αρχίσει και οριοθετήθηκε και μια συνοριακή γραμμή με τον γείτονα αυτόν. Είναι λοιπόν σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία χρειάστηκαν μάλιστα και σημαντικό πολιτικό θάρρος για να επιτευχθούν. Η σύσταση της Κομισιόν οδήγησε σε μια νέα εφορία του πληθυσμού υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν δημοσκοπήσεις που δείχνουν 96% μεταξύ των ε, κατοίκων της χώρας υπέρ της ένταξης. Άλλαξε λοιπόν το κλίμα πολύ από τα μέσα του 2008 όταν η ε, ε, Φιρόμ δεν μπόρεσε να μπει στην, ε, στο ΝΑΤΟ και που αυτό είχε οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και την Φιρόμ όπως, όπως υποστηρίζουμε την Κροατία. Υπάρχει από τη μία πλευρά ε, στη μία πλευρά, στη μία άκρη των Βαλκανίων η, ε, η ε, Κροατία και στην άλλη άκρη η Φιρόμ. Τώρα υπάρχει και η νέα ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει σημαντικές φιλοδοξίες για να συμβάλλει σε μια σταθεροποίηση των Βαλκανίων. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική όθηση που μπορεί να προσφέρει. Τώρα, η έκθεση θα πρέπει και αυτή να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και όσο δυνατόν ακριβέστερη. Νομίζω ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται τα πιο σημαντικά θέματα. Περιγράφω την, ε, τις πολιτικές εξελίξεις. Στην προσπάθεια συμμετέχουν όλο και περισσότερο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια συνολική εθνική προσέγγιση για την ένταξη. Είναι γνωστά βέβαια τα θέματα της διαφθοράς. Είμαστε ακόμα μακριά από μια τελική νίκη κατά της διαφθοράς. Αλλά έχει γίνει πιο αποτελεσματική προσπάθεια. Και η Βουλή έχει γίνει πιο αποτελεσματική. Καμιά φορά οι αποφάσει λαμβάνονται ίσω με υπερβολική ταχύτητα. Πάντω και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι από κάθε άποψη τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Οι εκλογέ που έγιναν την Άνοιξη, τοπικέ εκλογέ αλλά και προεδρικέ εκλογέ, απαιτέλεσαν σημαντικό βήμα πρόοδου. Δεν ήταν 100% όπως θα θέλαμε αλλά πάντως αποτελούν σημαντική πρόοδο απέναντι σε παλαιότερες εκλογέ. Πρέπει να τονιστεί ακόμα ότι η συμφωνία, η συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας εφαρμόζεται και ότι γίνεται προσπάθεια να αποφύγουν την χρήση προκλητικών συμβόλων ώστε να μην ανατρέψουν αυτή την ισορροπία που πάει να υπάρξει γιατί μιλώ και για αυτή τη λεγόμενη μακεδονική κυκλοπαίδεια η οποία έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ τους αλβανόφωνους. Το κράτος δικαίου ε, κάνει και αυτό βήματα πρόοδου. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι η πολυφωνία των μέσων. Τα μέσα είναι σε ιδιωτικά χέρια αλλά δεν, δεν υπάρχει επαρκής πολυφωνία. Η Μακεδονία πρέπει να κάνει και κάτι για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος μειονοτήτων και μιλώ κυρίως για τις γυναίκες. Είναι άσχημη η κατάσταση κυρίως των εργαζόμενων και κυρίως αυτών που εργάζονται στην υφαντουργία. Υπάρχει και υψηλή, υψηλό ποσοστό ανεργίας, αλλά Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι και στην οικονομική παραγωγή έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι. Και το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον έχει γίνει ελκυστικότερο. Σημαντικό για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός από αυτές τις διακοινωτικές σχέσεις μεταξύ των ε, εθνοτικών ομάδων δηλαδή, είναι και οι σχέσεις προς τους γείτονες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν ελαφρύνσεις στο καθεστώς των προξενικών θεωρήσεων που θα επιτρέψουν και μια καλύτερη διασύνδεση με την Ευρώπη. Είναι καλό που λύθηκαν τα προβλήματα, τα διμερή προβλήματα με το Κόσοβο. Στην πρώτη τελευταία και τελευταία παράγραφο θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους γείτονες, αλλά αυτά οδηγούν και σε διασπάσεις και μέσα στον ίδιο τον ε, πληθυσμό. Θα απευθύνω έκκληση σε όλες και όλους να έχουν, να είναι πιο ανεκτικοί ημένα απέναντι στους δε και να υπάρχει και περισσότερη αμοιβαία αναγνώριση. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη να τηρήσετε το δίλεπτο στις παρεμβάσεις σας. Διότι είμαστε περιορισμένοι χρονικά. Πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής για τις σχέσεις με το ΦΥΡΟΜ, ο κ. Χατζημαρκάκης. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ειδικά τα τελευταία που είπε δηλαδή που ζήτησε περισσότερη ανεκτικότητα και αλληλοκατανόηση, <clears throat> αποτελούν πολύ σημαντικά. Η έκθεσή του είναι ειλικρινή, αντικειμενική και ισορροπημένη. Και αυτά που είπε για μια antiquization είναι και αυτά σημαντικά. Είναι απαραίτητο να συγχαρούμε την κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που έχει εκπληρώσει σημαντικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή της πορεία. Είναι σημαντικό αυτό. Είπατε κι εσείς ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια ευφορία. Αλλά και με τη νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στην Ελλάδα, με τον Γιώργο Παπανδρέου, όλα αυτά οδηγούν σε μια πορεία που είναι καλό να προχωρήσει και <clears throat> να εκμεταλλευτούμε την όθηση αυτή που δίνεται. Τώρα, η πλήρης εφαρμογή της ε, Συμφωνίας της Οχρίδας. Μεγάλη σημασία για τις διακοινωτικές σχέσεις. Μίλησε για τις προκλήσεις που ενδέχεται να υπάρξουν ανάμεσα στι εθνοτικέ ομάδε, Μιλάει και για αυτέ τι παραγράφου του 6 και 19. Τώρα για τα θέματα του περιβάλλοντος. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία απασχολούν πολύ τον κόσμο εκεί μαζί με τι προξενικέ θεωρήσει. Οι, οι, οι λίμνες τους, τα ποτάμια του, είναι πάρα πολύ μολυσμένα και προκαλούν προβλήματα και στι γειτονικέ χώρε. Βρίσκω εδώ λοιπόν και κάτι που θα, ίσως θα ήταν καλό να αρχίσουν να λειτουργούν εκεί ευρωπαϊκά προγράμματα, έστω και πριν από την ένταξη. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ένταξης, τον Δεκέμβριο προβλέπεται συζήτηση. Νομίζω ότι ο εισηγητής αναφέρει αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ρήτρες διαφύλαξης, αλλά πρέπει να δώσουμε προοπτική, να δούμε δηλαδή τι ωφελεί τους ανθρώπους εκεί ελαφρύνσεις στο σύστημα των προξενικών θεωρήσεων, προγράμματα. Αυτά λοιπόν ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Τάλερ. Ευχαριστώ κύριε Χατζημαρκάκη. Για δύο λεπτά η κυρία Κοπά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο συνάδελφό μου τον Ζόραν Τάλερ για την έκθεσή του ε, στην οποία προσπάθησε να λάβει με μεγάλη ευαισθησία υπόψη όλα τα νέα δεδομένα στην περιοχή ε, η θέση της χώρας μου είναι σαφής και σε αυτό συμφωνεί η μεγάλη πλειοψηφία των, ευρωπαϊκών, ε, των πολιτικών κομμάτων ε, για το ποια πρέπει να είναι η λύση, ποια είναι η δική μας προτινόμενη λύση στην τελευταία διαφορά που μας ταλαιπωρεί. Παρόλα Παρ' όλα αυτά, ο νέος Πρωθυπουργό θέλει να δώσει μια νέα δυναμική στο διάλογο, έχει δεσμευτεί να προχωρήσει δυναμικά στην επίλυση αυτής της τελευταίας διαφοράς και τη θέση μας, τη θετική μας διάθεση απέναντι στη χώρα τη δείξαμε και με την απόλυτη, ε, με την απόλυτη τα καθαρή θέση στην ανάγκη για απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, όταν συζητήθηκε πρόσφατα. Τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι η περιοχή μας ακόμα υποφέρει από την εργαλειοποίηση της ιστορίας. Αυτή είναι μια παιδική ασθένεια. Στην Ελλάδα την περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Δυστυχώ ε, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία δεν έχουν απαλλαγεί ακόμα από αυτό το σύνδρομο γενικά το πρόβλημα στην περιοχή είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη και εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί όλο το επόμενο διάστημα γιατί αυτό δεν αφορά τη σχέση με την ελλάδα αφορά σίγουρα και τη σχέση με τη βουλγαρία και ίσω παράλληλα με τη, νέα διαδικασία τη νέα δυναμική διαδικασία για να βρούμε επιτέλου μια λύση στο χρονίζον πρόβλημα του ονόματο να πρέπει να υπάρξει και μια διαδικασία μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη που θα μπορεί να λύσει όλα τα άλλα θέματα που πραγματικά δηλητηριάζουν τι σχέσει ε, μεταξύ των κρατών τη περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κοπά. Η κυρία Γιαννακού έχει για δύο λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Τάλερ για την προσπάθεια που έκανε. Ε, η ε, πρόοδος που φαίνεται στην έκθεση βέβαια ε, υπάρχει σε αρκετά θέματα, αν και από την Επιτροπή τονίστηκε ότι ένα μεγάλο και σοβαρό ζήτημα που υπάρχει είναι η υπόθεση της διαφθοράς, η οποία και από τις δικές μου πληροφορίες δεν φαίνεται να προχωρεί καθόλου καλά στη γειτονική χώρα. Όσο αφορά στις διαφορές στην περιοχή, κύριε Πρόεδρε, επειδή πάρα πολύ έχει παρεξηγηθεί το ζήτημα αυτό που ανέκυψε με την Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια, και που υπάρχει μια συμφωνία στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών το επίσημο όνομα της χώρας να συμφωνηθεί με την Ελλάδα, δεν είναι θέμα ονόματος. Το θέμα του ονόματος είναι το σύμβολο. Ε, το θέμα αφορά κυρίως τη χρησιμοποίηση της ιστορίας με τον τρόπο που συμφέρει το σήμερα. Στη δημιουργία μιας εθνότητας που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον όχι γιατί η ελλάδα φοβάται τη γειτονική χώρα. Ε, η θέση των πολιτικών δυνάμεων στην ελλάδα είναι σαφής μπορεί να υπάρξει ένα σύνθετο όνομα για όλες τις χρήσεις και αυτή είναι μια υποχώρηση της ελλάδος σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. θέλω να υπενθυμίσω βεβαίως ότι όπως ακριβώς θεωρήθηκε για την κροατία ως benchmark η συμφωνία που έκανε με τη Σλοβενία και που ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν εις βάρος της Κροατίας, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κατανοηθεί ότι πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Δηλαδή τα κράτη-μέλη οφείλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους και η ένταξη χωρών που δεν θέλουν να λύσουν ορισμένα προβλήματα συναντά δυσκολίες και οφείλει να συναντά μια τέτοια συμπεριφορά την αντίθεση του συνόλου της Ευρώπης και όχι μόνο ορισμένων χωρών. Κατά τα άλλα κύριε Πρόεδρε, αν υπάρξει ανάγκη θα γίνουν σχετικές τροπολογίε, Θέλω και πάλι να συγχαρώ τον κύριο Τάλερ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Δύο λεπτά. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Τάλερ και του εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για την αντικειμενική και ε, ε ξεκάθαρη έκθεσή του. Ε, χαιρετίζω και τις πρόοδους που έχει κάνει η ΦΥΡΟΜ στην πορεία της προς μια ε, ένταξη και κυρίως στην οικονομία και στις κοινωνικές εξελίξεις. Υποστηρίζω και αυτά που είπε ο κύριος Μπροκ όταν λέει ότι οι νυν χώρες μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν ε, κολλήματα που, αξεπέραστα κολλήματα για την ένταξη νέων χωρών. Η στρατηγική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται και να ενισχύει μάλλον την περιφερειακή συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των γειτονικών χωρών. Και γι' αυτό υποστηρίζω και ελπίζω σύντομα η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας να λάβει μια ε, ημερομηνία ένταξη των, ε, ε, μάλλον των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ελπίζω να μπορούν να επιληθούν και τα προβλήματα που υπάρχουν με γειτονικέ της χώρες. Δεν μπορώ τώρα να πω και στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου τονίσαμε κατά επανάληψη ότι υπάρχουν τομείς που είναι ευαίσθητοι και προκλητικοί και για μας, τους Βουλγάρους αυτό το λεγόμενο hate speech που βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και μέσα στα σχολικά βιβλία. Εξακολουθεί και υπάρχει αυτό το κήρυγμα μίσους όπου ε, γίνονται και ορισμένε δηλώσεις απέναντι σε γειτονικέ χώρες που εν πάση περιπτώσει δεν θα μας άρεσε να παραμείνουν και στο μέλλον. Και θα χαρούμε ιδιαίτερα εάν μπορούν να γίνουν και κοινοί εορτασμοί για κοινά ε, ιστορικά γεγονότα με την ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της, Γερμανίας, της ε, Μακεδονίας και γι' αυτό έχω κάνει και ε, ορισμένες σχετικές τροπολογίες και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Κοβατσάκ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κύριλοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Πιστεύω και εγώ ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε με τις Ελπίζουμε όλοι οι γείτονε ότι με το θέμα των προξενιών θεωρήσεων θα βοηθηθούν κυρίως οι νέοι. Αυτό είναι κάτι που επιθυμούμε όλοι. Η όλη διαδικασία λοιπόν ένταξης θα έπρεπε να αρχίσει με την εξέταση της πραγματικής κατάστασης που σε αυτή τη χώρα για να βοηθηθεί η χώρα. Και εγώ συμφωνώ με την Ελληνίδα συνάδελφο, όταν βλέπω ποια είναι η διαδικασία για την ονομασία, το πρόβλημα δεν είναι η ονομασία ίσως, γιατί η Βουλγαρία πρώτα απ' όλα αναγνώρισε το συνταγματικό όνομα με την Φύρομ, ε, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Μίσος, ακραίες ε, εθνικιστικές τάσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να το λάβουμε υπόψη, διότι υπάρχει κλιμάκωση των εθνικιστικών τάσεων, κυρίως και εκ μέρους κυβέρνησης. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν ταχύτατα διαφορετικά. Και η Βουλγαρία έχει την εντύπωση ότι δημιουργείται ένα κλίμα μίσους στην ε, ε, χώρα αυτή που διαταράσουν το καλό κλίμα με τις γειτονικές χώρες. Στην παράγραφο 19 κάτι αναφέρεται και η αύξηση των εντάσεων με τους γείτονες είναι σημαντικό και θα πρέπει να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα ευθύς μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυρίλοφ. Για δύο λεπτά ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εμείς είμαστε υπέρ της έκθεσης Τάλερ. Ήμουν μέλος της ομάδας ε, φιλίας εγώ στην προηγούμενη Ελπίζω ότι θα μπορέσω να επισκεφθώ σύντομα την Μακεδονία και ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση Μακεδονίας για τις προσπάθειες που κάνει καταπολεμήσει την ε, διαφθορά και να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Σύντομα θα δω και τον Υπουργό Εξωτερικών. Πριν από ένα μήνα, στο Στρασβούργο δέχθηκα μία αντιπροσωπεία βουλευτών από τη χώρα αυτή και τους είπα να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους, και το επαναλαμβάνω τώρα, ότι δεν, και να το δηλώσουν δημοσίως, ότι δεν έχουν διάφορες ε, ε, εδαφικές διεκδικήσεις στις γειτονικές χώρες. Και θα ήθελα και το ΠΑΣΟΚ, η νέα κυβέρνηση της Ελλάδος, να μπορέσει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να επιληθεί το πρόβλημα την ονομασία, γιατί ώρες, ώρες είναι κομική αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα επίσης να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι λέγουν οι Έλληνες ότι στρατιωτικά μπορεί να τους απειλήσει το κράτος Μακεδονίας, όντας η Ελλάδα μέρος του ΝΑΤΟ. Τι να σας πω. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής θα γίνει αποδεκτή, θα το αποδεχθεί αυτό το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα βελτιώσει γενικότερα και τη σχέση μεταξύ της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Τάνο και για δύο λεπτά. Ο κύριος Πόσελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου Χατζημαρκάκη που πρόκειται από την πρώην γαλλική επαρχία του Σάρλαντ. Θα αναφερθώ και στον Ντανιέλ Κονμπέντιτ που είπε κάποτε ότι η Μακεδονία είναι η Μακεδονία είναι η Μακεδονία. Ας σταματήσουμε επιτέλους με τη, τα παιχνίδια αυτά με την ονομασία. Η Γαλλία λέγεται Γαλλία. Και δεν πάει επειδή ε, λέγεται France να ζητήσει να μπει στην Φραγκφούρτη. Η Γαλλικία λέγεται ε, Γαλλικία και στη Γαλλία, Γαλλικία και στην Ισπανία. Η Μεγάλη Βρετανία λέγεται Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν αξιώνει να πάρει ένα μέρος της Βρετάνης. Ας σταματήσουμε με αυτές τις ανοησίες επιτέλους. Αγαπητή Μαριέτα, σε αγαπώ και σε εκτιμώ, αλλά να λέτε ότι οι Μακεδόνες δεν υπάρχουν ως εθνική οντότητα, ε, δεν είναι πράγματα αυτά. Η μητέρα μου είναι Αυστριακή. Η, Αυστριακή, η Αυστρία, η Αυστρία για χίλια χρόνια ήταν έννοια υπερεθνική. Μόνο από το 1947 και μετά υπάρχει αυστριακό έθνος το οποίο αυτό αυστριακό έθνος. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Οι άνθρωποι μπορούν να αυτοαποκαλούνται όπως θέλουν. Εάν οι Μακεδόνες θέλουν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, ας μην έρθουμε εμείς εκ των έξω να αμφισβητήσουμε την ταυτότητά τους. Αυτά οδηγούν σε ε, ελλείψεις ισορροπιών. Και γι' αυτό χαίρομαι που ο κ. Στάλερ που δεν μιλάει για το παρελθόν. Ερχόμαστε εμείς τώρα στο Άχεν και δίνουμε το βραβείο του Καρλομάγνου και λέμε ότι αυτός ήταν ε, ο κοινό μας πατέρας. Ελπίζω κάποτε ε, να δοθεί και ένα βραβείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτός να είναι ο ιστορικός πατέρας όλης αυτής της περιοχής. Ο κύριος Αγκουράκης, εκτολόγια, δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συμβουλέψω τον προπροηγούμενο ε, εκπρόσωπο εδώ που μίλησε, τουλάχιστον όσον υπάρχει επίσημη ονομασία της χώρας αυτή να χρησιμοποιεί. Ε, ακούστηκαν διάφορα. Ε, δεν είναι σωστό ε, τη στιγμή που και στην έκθεση και γενικά μιλάμε για πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, ευρωβουλευτέ στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλάνε για Μακεδονία. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Διότι αυτό δεν βοηθάει στο να λυθεί το πρόβλημα. Το δεύτερο. Είναι αλήθεια και είναι γεγονός ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε και να κουραστούμε ακόμα περισσότερο ε, ή μάλλον πρέπει να κουραστούμε, γιατί δεν νομίζω το έχουμε κάνει, ώστε να επέλθει σταθερότητα, συνεργασία και ε, ε, φιλία στα Βαλκάνια. Φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγκρούονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έχουμε και τα ενεργειακά, έχουμε και τη Ρωσία, έχουμε και τους Αμερικανούς, έχουμε πολλά στην περιοχή. Οξύνονται αντιθέσει, οξύνονται τα προβλήματα. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα, συνεργασία και ασφάλεια. Για να τα πετύχουμε αυτά πρέπει να κινηθούμε βάσει αρχών και όχι βάσει τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, τι λέει η ιστορία τη μία χώρα και η ιστορία τη άλλη χώρα. Και εγώ μπορώ να απαντήσω στον κύριο από τη Γερμανία χιλιάδε άλλα ε, επιχειρήματα. Δεν είναι αυτό. Αυτό έγινε 20 χρόνια στα Βαλκάνια και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια διαδικασία υπό τον ΟΗΕ. Η έκθεση δεν κάνει καλά στο σημείο 19 που δεν αναφέρεται στη διαδικασία υπό τον ΟΗΕ για την επίλυση αυτού του ζητήματο, και με τον τρόπο αυτό δεν βοηθάει. Τέλο, δεν είναι θέμα ονόματο. Είναι θέμα συνόρων, είναι θέμα εθνικισμού, είναι τέτοια ζητήματα. Και τελειώνω λέγοντα το εξή θα χαιρόμουν πολύ περισσότερο εάν το ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει κάτι για το σημείο 14 όπου γίνεται λόγος για τα προβλήματα των εργαζομένων γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Διαπιστώσαμε στην έκθεση πρόοδου της Κομισιόν ότι η χώρα για την οποία μιλούμε, η χώρα με τις οποίες πρόκειται, έχει επιτελέσει σημαντικές πρόοδους. Και ότι αυτές οι πρόοδοι αποτελούν και τη βάση για να συζητήσουμε για ενδεχόμενη ενταξιακή πορεία. Θα αναθεωρήσω λίγο αυτά που είπε ο κ. Πόσελτ. Δηλαδή, συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει και από τις δύο πλευρές. Να μην εγερθεί εντύπωση ότι ενισχύεται η μία πλευρά με ομιλίες που κάνουμε εδώ τόσο πολύ ώστε να μην έχει πια διάθεση να προχωρήσει σε συμβασμό με την άλλη πλευρά. Πόσελτ δεν είναι Γαλλία, είναι Γαλλική Δημοκρατία. Δεν το λέει κανένας έτσι όμως βέβαια. Επιβλή Φρανσέζ. Άρα θα μπορούσε να ε, δοθεί η σύσταση στην μακεδονική κυβέρνηση να δεχθεί το μακρότερο δυνατό όνομα. Το πιο μακροσκελές. Όσο μακροσκελέστερο είναι το όνομα αυτό, τόσο περισσότερο θα έχουμε και εμείς αφορμή για να ε, λέμε μόνο Μακεδονία. Και με χώρα μου λέγεται Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για να μην λέμε όλο αυτό το μακρινάρι, λέμε Γερμανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε το θέμα με τρόπο ανεκτό για όλους. Και ε, στην Ελλάδα δεν είναι θέμα τώρα ε, των λίγων εθνικιστών, είναι δημοκράτες και ε, σοσιαλδημοκράτες. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αν θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε τώρα για τον Μεγαλέξανδρο στην Ελλάδα ή αν θα πρέπει να περιμένουμε ε, λίγο και ε, ίσως δεν είναι και απαραίτητο στους επίσημους επισκέπτες να προσφέρεται η νεκρική μάσκα του Μεγαλέξανδρου. Ίσως μπορούμε να περιμένουμε λίγο να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, ώστε να μπορέσουν και σύντομα να αναβληθούν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Για δύο λεπτά το λόγο τον έχει η συνάδελφος κυρία Λούνατσεκ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα για την ονομασία, για την χώρα για την οποία εδώ μιλούμε. Να κάνω και εγώ λίγες παρατηρήσεις. Ως πολίτης μιας χώρας η οποία όντως θέσπισε και ονόμασε την ταυτότητά της εδώ και λίγες δεκαετίες και πριν από τον δεύτερο πόλεμο ορισμένοι έλεγαν ότι η Αυστρία είναι ξεχωριστή χώρα. Μην ανησυχείτε κύριε Πόσελτ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα της ταυτότητας εξακολουθεί να είναι τέτοιο που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Και στη δική μου χώρα την Αυστρία το ίδιο. Χρειάστηκε χρόνος μέχρι ότου πολλοί να αποδεχθούν ότι έχουμε και εμείς οι ίδιοι αυτή την ταυτότητα. Αυτό που δεν κατανοώ πραγματικά είναι σε ορισμένες Ελληνίδες και Έλληνες έχω την εντύπωση ότι έχουν τον μεγάλο φόβο ότι η χώρα τους, το κράτος τους, η Ελλάδα, που είναι και έχει μια ε, ιστορική ταυτότητα, παγκόσμια γνωστή, έχει το φόβο τώρα ότι θα του ε, τους προκαλέσει κάποιο πρόβλημα μια μικρή χώρα που βρίσκεται στα βόρεια σύνορά τους. Όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ προηγουμένως, θεωρώ ότι η μακεδονική κυβέρνηση θα πρέπει και αυτή βέβαια να προσέξει πολύ το ύφος τη ρητορική που ασκεί, να μειώσει λίγο τις εντάσεις και να αποφύγει τα εθνικιστικά. Αυτό θα ενισχύσει και τις προσπάθειες που καταβάλλονται τώρα από την ελληνική πλευρά και όπου έχουμε εμπιστοσύνη, όπω είπε και η κυρία Κοπά, στι προσπάθειε τη νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, βρίσκω την έκθεση Τάλερ σε πολλά θετική. Ένα βρίσκω πολύ σημαντικό και θα πρέπει να περιληφθεί. Ήδη πέρυσι, στο τελευταίο ψήφισμά μα, έλεγε ότι τα διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να αποτελέσουν κόλλημα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και στην έκθεση του κ. Αλμπερτίνη, του Προέδρου, έχουμε μια σχετική παράγραφο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να περιληφθεί και στη δική σας. Και τέλος για τις παραγράφους 15 και 16, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στις δημόσιες συγκοινωνίες και όχι μόνο οι μακεδονικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελεί σημαντική δυνατότητα που διευκολύνει τη μετακίνηση των ανθρώπων και χρειάζονται προσπάθειες εκατέρωθεν. Σας ευχαριστώ κυρία Λούνα Τσεκ. Ολοκληρώνει τη συζήτηση ο κ. Κουμουρτζάκος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν είναι το θέμα της σημερινή συζήτησης αλλά μια κρινόμενη για, ένταξη, για την ενταξιακή της πορεία χώρα η ιστορία κύριε πρόεδρε δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για το παρόν και το μέλλον και σε αυτό θα συμφωνήσω με όσους έχουν μιλήσει αλλά όταν η ιστορία αγνοείται ειδικά στα βαλκάνια μπορεί να επιστρέψει με το χειρότερο πρόσωπό της ειδικά όσον αφορά στην έκθεση στην πρόταση ψηφίσματος. Ορθώς επισημαίνεται στο ψήφισμα μια αξιοπρόσεκτη πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του πολιτεύματος της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης στην πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως παραδείγματο χάρη η ικανοποιητική σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών. Ταυτόχρονα όμως το υποσυζήτηση ψήφισμα διακρίνεται από μια τάση υπερβολικής, θα έλεγα, ωρεοποίησης της κατάστασης στην χώρα αυτή. Υποβαθμίζονται τα μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, την εκτεταμένη διαφθορά, τις εθνοτικές σχέσεις. Υποβαθμίζεται επίσης και θα έλεγα ότι αγνοεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση Γκρουεύσκη σταθερά υιοθετεί έναν ακραία εθνικιστικό, μυσαλόδοξο και επιθετικό λόγο. Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε κύριε Πρόεδρε το γεγονός ότι η εθνικιστική αυτή ρητορία αλλά και συγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης Γκρουεύσκη έχουν δημιουργήσει τριβές με δύο γειτονικές της χώρες που και οι δύο είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία και η Ελλάδα ο σεβασμό είχα τη δυνατότητα και σα ευχαριστώ γι' αυτό να το αναφέρω και χθε ότι ο σεβασμό τη αρχή τη Καλή γειτονία είναι θεμελιώδου σημασία για την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα αλλά και για κάθε πρόοδο στην ευρωπαϊκή προοπτική των ενδιαφερομένων για ένταξη χωρών. Η εξέβριση μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα τη ονομασία στην τρέχουσα διαδικασία διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ είναι πράγματι κομβική σημασία. Άλλωστε, πρόκειται να γίνει μια νέα συνάντηση στι 16 Νοεμβρίου είναι κομβική σημασία για να υπάρξει συνέχεια, στη συνέχεια πρόοδο προ την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Για όλου αυτού του λόγου θα κατατεθούν σχετικές τροπολογίες στο υποσυζήτηση ψήφισμα. Και μια τελευταία αναφορά, κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα του ονόματος δεν είναι απλό. Μιλάμε για μια περιοχή που λέγεται Μακεδονία, τμήματα της οποίας ανήκουν στην Ελλάδα, τη χώρα μου, τη Βουλγαρία και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουμε μία περιοχή, τρεις χώρες, τρεις λαούς. Δεν μπορεί ένας να έχει το όνομα και να έχει το μονοπόλιο του ονόματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Και τώρα η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Αλεξάνδρα Χράγχε, έχει το λόγο ίσως για παραπάνω από τρία-τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιε παρατηρήσει θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι είναι πολύ ισοσκελισμένη και καλά ενημερωμένη συζήτηση. Επίσης ισοσκελισμένη είναι και η έκθεση και η Επιτροπή γενικά συμφωνεί με το περιεχόμενό της. Τώρα, αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό για αυτή τη χώρα στο επόμενα χρόνια είναι δεδομένου ότι έχουμε ένα κοινό στόχο να αρχίσουν οι διαδραματέσεις. Ποια είναι λοιπόν η σύστασή μας, επειδή πιστεύουμε ότι, είναι, ότι πληρούνται επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια να προχωρήσουμε. Πού θα μπορούσαμε να κάνουμε λάθος ε, στην στρατηγική μας, στις μεταρρυθμίσεις. Μιλώντας για μεταρρυθμίσεις, θα ήθελα να μιλήσω για το εξής θα πρέπει να υπάρξει γενικότερη μεταρρύθμιση όλου του πλαισίου του ρυθμιστικού και του διοικητικού της χώρας αυτής πριν να αρχίσουμε τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Πού θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Το όνομα του ονόματος. Όσο και ανόητο αν φέρεται σε κάποιον μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρόσκομα. Έχουμε λοιπόν εδώ μία μοναδική ευκαιρία και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την χώρα αυτή να επιλύσει το πρόβλημα της ονομασίας της στο εγκύτατο μέλλον. Διαφορετικά αυτό το οποίο διακινδυνεύουμε, συγγνώμη, να μην ανοίξει ποτέ διαπραγματεύσεις. Οποιαδήποτε λοιπόν συμφωνία θα είναι καλή. Και νομίζω ότι πρέπει εδώ να υπάρχει πολιτική δέσμευση όχι μόνο ημών και του ΟΗΕ αλλά και σε υψηλότητα το επίπεδο της χώρας αυτής. Συμπερασματικά. Πού πάμε με τη Μακεδονία. Τέλος πάντων αυτή τη χώρα διορθώνει η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μέλλον στο πρόβλημα με αυτή τη χώρα και θα μείνει εκτό η Μακεδονία, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσουμε πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά, αυτές τις Για να ολοκληρώσει και ο στάλερ και ελπίζω αυτές οι, οι παρεμβάσεις να είναι σύντομε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους συζήτησαν το θέμα. Όλοι συνειδητοποιούμε ποιες είναι οι ευθύνες μας και ότι είναι αναγκαίο να προοδεύσει στο εγγύς μέλλον η Μακεδονία. Εμείς έχουμε λάβει δεσμεύσεις για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Και συμφωνώ. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι άμεση επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο για να επιληθεί το θέμα της ονομασίας. Πρόκειται για την πρώτη προτεραιότητα. Και θα πρέπει να βάλουμε στο ίδιο τρένο με την Ισλανδία και τη Μακεδονία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε με καλή συνεργασία να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Πραγματικά σύντομο. Ο Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 9 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή μεταξύ 25 και 28 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ρία Όμεν Ρόιτεν και στην οποία δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, αν μπορείτε παρακαλώ. Ja, voorzitter, eh, veel dank. Voorzitter, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ως εισηγήτρια τους επόμενους μήνες θα παρακολουθήσω εκ του σύναγγης τον τόσο σημαντικό αυτό φάκελο με αντικειμενικό τρόπο. Το μήνυμα στην Τουρκία πρέπει να περάσει υπό μορφή συστάσεων που θα υποβάλει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου στη χώρα αυτή. Και θα ήθελα με όλους τους συναδέλφους την καλύτερη δυνατή συνεργασία ώστε να υπάρξει βέλτιστη υποστήριξη. Στην έκθεση για την Τουρκία υπάρχουν δύο θέματα που επανέρχονται κάθε χρόνο. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία μπλοκάρουν οποιαδήποτε πρόοδο και πρέπει να πω ότι λείπει και δυναμική διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Τα πάντα φτάνουν μπροστά από το συνταγματικό δικαστήριο και καταραίουν. όπου και αν προβλέπονται μεταρρυθμίσει στο Σύνταγμα ή σε, άλλου, σε άλλα νομοσχέδια, σε άλλους νόμους, φερειπίν σε άλλου τομεί. και θα μιλήσω, θα αναφέρω ω παράδειγμα τον νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, στη θεωρία ο νόμος είναι πολύ καλός, αλλά στην εφαρμογή δεν γίνεται τίποτα. Βλέπουμε στα χωριά, στα μικρά αστυνομικά τμήματα, να υπάρχει άγνοια, να μην κάνει κανείς αυτό που πρέπει να κάνει και θα ήθελα στην έκθεσή μου να τα αναφέρω αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλω γραπτό σχέδιο ψηφίσματος και όπως είπα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δικαιοσύνη στην Τουρκία είναι ανεξάρτητη, πολύ ανεξάρτητη. Δεν είναι όμως αμερόληπτη και πιστεύω ότι η στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον δικαστικό τομέα για να μπορέσει να είναι επιτυχής θα πρέπει και τύπης και επί την ουσίας να γίνει από, το τουρκικό, από την τουρκική βουλή χωρίς μικρά κόμματα να μπλοκάρουν την όλη διαδικασία. Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα πρέπει να μπορεί κανείς να στηρίζεται στην δικαιοσύνη η οποία πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα και αμερόληπτα. Επίσης πρέπει να πω ότι κάποιοι νόμοι εγκρίνονται, περνούν και δεν εφαρμόζονται. Το ίδιο σημαίνει, συμβαίνει και για θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες. Σε κάποιες ε, ε, προσφυγές στη δικαιοσύνη δικαιώθηκε μια γυναίκα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ η απόφαση του δικαστηρίου. Η εκ της, ε, η καταχρηστική εξουσία της ε, αστυνομίας ε, είναι μεγάλη, κυρίως κατά των συνδικαλιστικών οργάνων και πάντα υπάρχει το πρόβλημα ότι πολλά πράγματα σκοντάφτουν μπροστά από το συνταγματικό δικαστήριο. Δεν είναι λοιπόν συνεκτικά αυτά με μια μοντέρνα κοινωνία στην Τουρκία που θα έπρεπε με δημιουργικότητα να προχωρήσει. Επίσης το θέμα της ε, ανεξιθρικίας, της θρησκείας, συγγνώμη, το δικαίωμα να μπορεί κανείς ε, να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του πιστεύω. Υπάρχει εξωτερική πολιτική, Υπάρχει το θέμα της ε, διαφθοράς. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι θετικός. Μεν. Και όταν ο Ερντογάν πηγαίνει στην, ε, στο Ιράν, στην Τεχεράνη και δεν λέει τίποτα για τα πυρηνικά δεν είναι στο ίδιο μήκο κύματο με την Ευρώπη. Επίση, υπάρχει το πρόβλημα τη Κύπρου. Η Τουρκία Μήπως μπορείτε κάπως να ηρεμήσετε στην αίθουσα, λέει κάποιος, για το συμπληρωματικό πρωτόκολλο δεν μπόρεσε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε κάποια θετικά μηνύματα και συμφωνώ με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ο κύριος Πάτσης είναι εξαιρετικός διαπραγματευτής, αλλά υπάρχει και το άνοιγμα προς τους Κούρδους. Εδώ και πέντε χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ακολουθήσει αυτή την τάση το Κοινοβούλιο. Κάποιος είπε στην Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η τουρκική κοινωνία είναι πιο σύγχρονη από αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, κυρία Μενράιτερ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχετε υποβάλει γραπτό κείμενο. Δεδομένου ότι Προβλέπετε συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης με 3 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. το τώρα ένα λεπτό που θα θεωρηθούν ως εισαγωγικές. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των αγοριτών. Μπρίπολς, Μάτλενερ, Τιοκάρους, Τάνοκ, Τάνοκ Βάιγελ Stop, ο κύριος Οβιόλς πρώτα απ' όλα. Για δύο λεπτά. Εάν τα λόγια της συναδέλφου συμφωνούν με το σχέδιο ψηφίσματος που θα μας υποβάλει, νομίζω, πράγμα το οποίο δεν αμφιβάλλω, μου φαίνεται ότι μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ευρύτατη συμφωνία για την έκθεση αυτή. Τρει πάρα πολύ σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα θετικό αλλά αυστηρό συγχρόνω. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές πολιτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών ή τεχνητά εμπόδια. Δεύτερον, η Τουρκία έχει αναλάβει σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να και να βοηθήσουμε αλλά και να απαιτήσουμε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Επίσης, το θέμα της Κύπρου, για να σταματήσει αυτός ο χωρισμός στα δύο της Κύπρου θα πρέπει να επιληθεί. Επίσης, έχουμε την εντύπωση ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουμε και κάποια εναλλακτική λύση στις δικές μας ε, τις ε, σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να επικαλεστούμε στο μέλλον. Πάκτα σουν σερβάντα. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο και ο Χάουιτ. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μανουράιτορ. Την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε μαζί στην Άγκυρα και ως κοινοβούλιο είδαμε περί των σπρόκειται και συμφωνούμε ότι θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί όλα τα μέλη της Επιτροπής που πήγαμε εκεί συνεισφέραμε, όντως αναγνωρίσαμε ότι ε, υπάρχει πρόοδος αλλά υπάρχουν και κάποιες τροχοπέδες. Δεν θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πούμε ότι έγιναν σημαντικά βήματα με τους Κούρδους, με το θέμα των σχέσεων με την Αρμενία, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ ε, αποφασιστική και σκληρή για να μπορέσουν να επιτευχθούν διάφορες συνταγματικέ μεταρρυθμίσει. Βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλέ επικρίσεις για την Τουρκία, το βλέπουμε αυτό στα πλαίσια της διεύρυνσης και θα θέλαμε το πρωτόκολλο της Άγκυρας να μπορέσει να εγκριθεί. Πιστεύω όμως ότι όλοι κάνουμε επικρίσεις. Δεν θα εισακουστούν οι πολύ αυστηρέ επικρίσεις θα πρέπει να, οι κρίσει μας να ακουστούν επικοδομητικά και να επενέσουμε τις προόδου που γίνονται. Όπως λέει η κυρία Ομενρόιτεν ότι η τουρκική κοινή γνώμη ε, θέλει να, ε, να μπει στην Ευρώπη. Αυτοί νομίζουν ότι δεν τους θέλουμε έχει σημασία ο τρόπο με τον οποίο του μιλάμε για να σχηματίσουν ε, εικόνα για μας. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει το κείμενο, οπότε σήμερα είναι προκατατικές απόψει που ακούγονται. Η πραγματική συζήτηση θα γίνει αρχέ Δεκεμβρίου. Από την 1η μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου θα είναι έτοιμα τα κείμενα. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνετε εδώ στο ένα λεπτού για κάποιε προκατατικές παρατηρήσει. Ο κ. Μαυρονικόλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ορθές οι παρατηρήσεις που ακούστηκαν από όλους τους προηγούμενους ομιλητές. Εκείνο το οποίο πρέπει και οφείλουμε να αναφέρουμε είναι ότι η Τουρκία όντως έχει πολλά προβλήματα. Αναφερόμαστε σε προβλήματα στο εσωτερικό και αναφερόμαστε στο αρμενικό, το κουρδικό και το κυπριακό πρόβλημα. Και αν δεχόμαστε ότι στην πράξη έχει γίνει μια προσπάθεια σε σχέση με το κουρδικό, αναμένει κανείς ότι και η Τουρκία δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς κάποια προσπάθεια το κυπριακό πρόβλημα. Και αναμφίβολα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υλοποιήσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας πρώτον, δεύτερον να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον να βοηθήσει ουσιαστικά στις συνομιλίες για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Εάν η Τουρκία έχει την καλή διάθεση, τότε μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα για το κυπριακό πρόβλημα. Και αυτό πιστεύω ότι θα ωφελέσει και την ίδια για την πορεία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρονικόλα. Ο κύριος Πρέμπολς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η κυρία Πρέμπολς, μάλλον, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Όμεν Ρόιτεν για τα αρχικά της σχόλια και υποστηρίζω τη γενική της γραμμή και τις προτεραιότητές της. Θα ήθελα όμως να προσέξει όλος ιδιαιτέρως την πρώτη αυτή πρωτοβουλία για τους Κούρδους. Πάντα ζητούσα να προσέξουμε το θέμα ιδιαίτερος. Πολλά πρέπει να γίνουν εκεί. Ναι, είναι ένα θετικό μήνυμα που βγαίνει, αλλά για την ώρα δεν είναι καθόλου καθαρό τι πρόγραμμα είναι αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τι λεπτομέρειε τη πρωτοβουλία αυτή. Απλώς λέει ότι πρακτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν και φοβούμε ότι αυτό ίσως να είναι απλώ μια τουρκική λύση, καθαρά τουρκική λύση. Δεν υπάρχει πραγματικό διάλογο με εκπροσώπου των Κούρδων σε αυτή τη φάση. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια προπόθεση. εάν θέλουμε να πετύχουμε μια καλή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πέραν από αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά αρνητική όσον αφορά τι πρωτοβουλίε που έχουν δρομολογηθεί μέχρι τώρα, σχετικά με τους Κούρδους, σχετικά με τους περιορισμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, περιορισμού στην παιδεία, τη χρήση των γλωσσών, ε, και όλα αυτά. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά αργότερα και να συμπεριληφθεί αυτή η σύσταση στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά θα δούμε θα γίνει. Παρακαλώ για ένα λεπτό επόμενη. Ο κύριο επόμενος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία όταν αποκαλείται φίλος του Ιράν. Είναι αλήθεια ότι είπε ο Ερντογάν ότι το Ιράν είναι ο μεγάλος φίλος της Τουρκίας. Έτσι φαίνεται. Το Ιράν που θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ από το χάρτη, που θέλει να έχει πυρηνικό πλεισμό, το Ιράν του Εσμπολά, τον, ε, και ο μεγάλος χώρος της Δύσης, μέγας φίλος της Τουρκίας. Και τι θέλουμε τώρα, να ε, διαπραγματευτούμε με αυτή τη χώρα. έχει βάλει εδώ και τόσα χρόνια και καταλάβει τη μισή Κύπρο και θέλετε να διαπραγματευτείτε μαζί τους. Τι θέλετε. Είμαστε με τα καλά μας. Να μιλήσετε για πάρα πολύ σοβαρέ κυρώσει κύριε και να μην καλλιεργείτε αυτό το φιλικό κλίμα τους Τούρκους διότι οι Τούρκοι μα κοροϊδεύουν και το μόνο το οποίο μπορώ να σκεφτώ για να βελτιωθούν τα πράγματα είναι να διακοπούν αμέσω οι διαπραγματεύσει. Για ένα λεπτό, κύριε Στάνοκ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω δύο θέματα. Κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα μου έθεσε κάποιος από την εκλογική μου περιφέρεια στο Λονδίνο, που μου λέει η Επιτροπή χορήγησε σημαντικά κονδύλια για την βελτίωση των δικαιωμάτων των ζώων στην Τουρκία. Διότι φαίνεται ότι τα μεταχειρίζονται και στον αγροτικό τομέα και αλλού. Είναι αλήθεια αυτό. Κάνει κάτι, ξέρει τόσο καλά την κατάσταση και κάνει κάτι για να του βοηθήσει. του ε, Τούρκους για τα, αυτό που κάνουν οι επιτροποί. Δεύτερον, Ξέρουμε ότι υπεγράφει πρωτόκολλο μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας και την επομένη είπε δημοσίως ο Πρωθυπουργό ότι ποτέ δεν θα κυρωθεί η συμφωνία αυτή εκτός εάν επιληθεί εκ των προτέρων το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και έτσι είπε ότι εμείς ποτέ θα το περάσουμε στη Βουλή, θα το υποβάλουμε στη Βουλή προσκύρωση κυβέρνηση της Αρμενίας επέδειξε εξαιρετικά μεγάλη πολιτική βούληση για να επιληθεί αυτό το θέμα και, και η διασπορά παντού κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντική ήταν η συμβολή και η καλή θέληση της Αρμενίας για να μπορέσει να επιδευτεί αυτή η Τουρκία. Ευχαριστώ. Ο το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ για πολλωστή φορά θέλω να πω ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται και τη συμφέρει να έχει δίπλα της μια Τουρκία εκδημοκρατισμένη που να σέβεται τους γείτονες της. Και βεβαίως δεν λέμε κάτι υπερβολικό και καταλαβαίνω ότι πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μας βλέπουν ως μονοθεματικούς εδώ, να ασχολούμαστε δηλαδή συνεχώς μόνο με το Κυπριακό, αλλά τι θα κάνατε εσείς εάν ένας γίγαντας δίπλα από τη χώρα σας καταλάμβανε τη μισή σας χώρα. Να πάψει η Τουρκία να κρύβεται πια πίσω από το τι έκαμε το 2004. Να ενεργήσει με προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τέτοιες που να συνάδουν με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και προς την κατεύθυνση μιας λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία ηθαγένεια, μία διεθνή κυριαρχία, μία προσωπικότητα. Αυτό αν το κάνει εμείς είμαστε μαζί της. Σας ευχαριστώ. Θεοχάρους το επόμενο όνομα, κύριε Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Θεοχάρους, συγγνώμη. Όλοι οχυρώνονται πίσω από τη θέση ότι διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίε στην Κύπρο. Η Τουρκία αυτό κάνει. Όσοι από εμά δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα, αυτό κάνουν. Και η Τουρκία δεν εκπληρώνει καμία από τι υποχρεώσει τη. Κανεί δεν μπορεί να μα διαβεβαιώσει ότι οι συνομιλίε αυτέ πάνε καλά. Και πρέπει να ξέρετε ότι δεν πάνε καλά. Οδηγούνται προ μια τουρκική λύση, όπω ελέγχθηκε προηγουμένω για το κουρδικό. Γιατί μόνο αν δεχθούμε τι τουρκικέ θέσει θα ε, υπάρξει μια συμφωνία. Αν διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μα, θα ε, μένουν πάντα στη γωνία. Πρόσφατα ο κύριος Σταλάτ πριν δύο μέρες είπε, ο εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων είπε ότι το εδαφικό ένα ακαθόδες πρόβλημα της Κύπρου, θα, του κυπριακού προβλήματος θα επιληθεί με την με τον σχεδιασμό των συνόρων μεταξύ των δύο κρατών. Αυτό είναι το ενίο κράτο που θέλουν να εφαρμόσουν στην Κύπρο. Και θα μετακινηθούν, λέει, 50.000 Τουρκοκύπροι. Δεν είναι Τουρκοκύπροι που θα μετακινηθούν, είναι έπικοι, γιατί οι Τουρκοκύπροι διάλεξαν πολύ καλά σε ποια σημεία εγκαταστάθησαν, γνωρίζοντας ποια ενδεχομένως κομμάτια θα επιστραφούν. Εμείς ζητάμε από την Τουρκία να επιστρέψει πάρα αυτά την πόλη τη Αμοχώστου του ως ένα δείγμα καλή θέληση αν θέλει να στηρίξει τι συνομιλίε και η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που θα υποχρεώσουν την τουρκία να έρθει με λογικές προτάσεις στις συνομιλίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Θεοχάρου. Τέλει, ο κύριος Βάιγκελ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Eh, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ δηλαδή με τα πρόσωπα εκείνα που θεωρούν την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ε, μελλοντική χώρα μέλος. Άλλωστε, πρέπει να δουν υπόψη και ιδιαίτερε ευαισθησίε τη Τουρκία και να αντιμετωπιστούν με καλή θέληση. Είναι καλό να αναφέρουμε τι προοδού στου διαφόρου τομεί. και βέβαια για την τήρηση τον κ. της αλλά και για, για το γενικότερο κλίμα στην Τουρκία και απέναντι στις μειονότητε και απέναντι στον τύπο. Από την Τουρκία αναμένουμε κάπως περισσότερη δέσμευση για το Κυπριακό, για τη λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία θα πρέπει να αποσύρει ένα μέρος των δυνάμεων τουλάχιστον ω δείγμα καλής Η Τουρκία έχει ζητήσει μάλιστα να συμμετάσχει σε διάφορε ειρηνευτικέ αποστολέ με δυνάμει και μάλιστα ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Άρα θα μπορούσε να κάνει και αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την ακούμε γιατί συζητούμε το κείμενο που μας έδωσε η συγγήτρια. Μπορεί να σχολιάσει συντομότατα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Ακούσα τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων και θα προσπαθήσω στα πλαίσια του δυνατού να λάβω υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί και από την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων η έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Ωραιότατα, ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, των επόμενων βημάτων, όπως είπαμε, αρχές Δεκεμβρίου θα υπάρχει το κείμενο και συζήτηση του κειμένου που 1 μέχρι 3 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Από 26 ως 27 Ιανουαρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και προβλέπεται το Φεβρουάριο ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Περιμένουμε τον Υπουργό κύριο Γέρεμικ, Βουκ Γέρεμικ, Λοιπόν, δημιουργία ενός οικονομικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες, τροποποίηση του κανονισμού. Γνωμοδότηση της εισηγήτριας της κυρίας Μπάρμπαρα Λόκμπίλερ, που έχει το δικαίωμα να παρέμβει. Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το συζητάμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα το θέμα, οπότε θα εστιαστούμε στη νομική βάση του μέσου. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 181α σαν την αποκλειστική και μοναδική νομική βάση. Μέχρι τη ότου τεθεί σε ισχύ η Λισαβόνα αυτό το άρθρο δεν δίνει νομοθετική εξουσία στο Κοινοβούλιο. Μετά από τη Λισαβόνα η συναπόφαση θα είναι η συνθισμένη διαδικασία. Στην πρώτη συνάντηση με τον Χέλμοντ Σόλτ, με τον εισηγητή, φαίνεται ότι συμφωνούμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν υιοθετηθεί η έκθεση μετά από την θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο εισηγητή ετοίμασε μια, ένα πρώτο σχέδιο εκθέσεως που θα συζητηθεί ε, στις 10 ε, Νοεμβρίου. Ο κ. Σόλτ συμφωνεί στην πρότασή του με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί ο κανονισμό μόνο στο άρθρο 181α, ε, το οποίο στερεί από το Κοινοβούλιο τι εξουσίε του όσον αφορά τη συναπόφαση. τα περισσότερα άλλα μέσα τη εξωτερική σχέση χρησιμοποιούν τη διτή νομική βάση, το 181α και το 179 όπω η πολιτική η γειτονία στα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέσο για τη σταθερότητα. Στη συνθήκη της Λισαβόνα ε, έχει προσθεθεί μια εξήγηση στο άρθρο 181α, επεξήγηση, που θα γίνει άρθρο 212 το 181α. Εκεί ρητά περιορίζεται η συνεργασία στα πλαίσια του άρθρου αυτού σε τρίτες χώρες εκτός των ανεπτυγμένων, των ανεπτυγμένων χωρών. Συγγνώμη. Και δημιουργείται αμφιβολία κατά πόσο η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστηρίζεται από τον συγκητή Τσίντα αρκούν ω νομική βάση για τη συνεργασία και μέτρα συνεργασία με αναπτυσσόμενε χώρε. Εγώ θα πρότεινα αυτό το θέμα να παρουσιαστεί στην Νομική Επιτροπή για νομική εξέταση σύμφωνα με τη διάταξη 37 του εσωτερικού κανονισμού. Και άλλη πρόταση που κάνω είναι ήδη να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να προβεί σε μια αξιολόγηση της καταστάσεως μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης εφόσον μόλις δύο μήνες απομένουν μέχρι μια νέα συνθήκη θα πρέπει να ξέρει το Κοινοβούλιο επακριβώς ποια είναι η διαφορά μεταξύ υιοθετήσεως του κανονισμού στα πλαίσια της Νίκαιας ή της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Ίντα κανονικά θα πρέπει να περιμένει μέχρι ότου ληφθούν και άλλα βήματα για υιοθέτηση. Μάλλον να περιμένει μέχρι να τοποθετηθεί η νομική βηματα για υιοθετηση μαλλον να περιμενει μεχρι να τοποθετηθει νομικη υπηρεσια και η νομική επιτροπή. Και μετά θα συζητήσουμε ε, μέσα σε ένα κοινό συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα και θα σταματήσω εδώ πέρα διότι μου υποσχεθήκατε ότι θα συζητήσουμε αυτό το μέσο περαιτέρω στην επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα, λέει ο Πρόεδρος, να μην δώσω το λόγο και στον συζητητή. Νομίζω ότι τα συνοψίσατε όλα. Παρακαλώ, μην κάνετε ιδιωτικέ συζητήσει εδώ, αλλά έξω εφόσον συνεχίζετε η συνεδρίαση ή να καθίσετε ήσυχα. Κύριε Γκάλερ, για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω. Μήπως μπορείτε να είστε πιο ήσυχοι. Είτε ψυγείστε είτε βγείτε έξω. Υποστηρίζω τα όσα είπε η κυρία Λόχμπιλερ. Έχουμε το πρόβλημα ότι για τη συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς όπου ε, δεν μπαίνουν σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Και γι' αυτό είναι σωστό να προσαρμοστεί το ICI. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα, αφενός, με τη νομική βάση που προτείνει ο εισηγητής της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, κάτι το οποίο ε, αποτρέπει, δηλαδή δεν επιτρέπει μάλλον την συναπόφαση και από την άλλη μεριά με το άρθρο 212 υπάρχει το μέγα πρόβλημα ότι το άρθρο αυτό λέει συνεργασία με τρίτες μη αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ αυτό που θέλουμε είναι, στην πραγματικότητα, είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολιτικές σε συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες και εκτός της ε, ενίσχυσης στην ανάπτυξη. Ε, ε, και δεν το πετυχαίνουμε έτσι και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσουμε νομικές συμβουλές όπως είπε και η εισηγήτρια και η Κομισιόν. Ούτως ή άλλως ο μηχανισμός θα πρέπει να μετονομαστεί και να λέγεται ε, μηχανισμός συνεργασίας με χώρες μη ODA. Αν εξετάσουμε όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο, θα δούμε ότι, εδώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια, ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα και από κάπου πρέπει να εξευρεθούν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι εάν μεταφέρουμε κάποια καθήκοντα σε ένα νέο μηχανισμό, πρέπει να μεταφερθούν και οι πιστώσει, τα κονδύλια. Εάν ε, και επειδή δεν θα έχουμε νέα χρήματα, νομίζω ότι θα πρέπει για να είμαστε συνεπεί να τα πάρουμε από τον DCI. Βέβαια, αυτό είναι η συζήτηση επί της ουσίας, που δεν έχει άμεση σχέση με την νομική βάση. Πάντως, θέτω υπόψη σας τον προβληματισμό αυτό. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας κύριε Γκάλερ. Όπως ζήτησε η συγγήτρια, η νομική υπηρεσία θα γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνο, ούτως ώστε την επόμενη συνεδρίαση να, στις 10 Νοεμβρίου να έχουμε αυτή τη γνώμη. Πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά θα ακούσουμε τον Υπουργό τον κύριο Βουκ Γέρεμικ.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 Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε, διότι είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση που την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας. Σας παρακαλώ συνάδελφοι να καθίσετε. Όποιος ενδιαφέρεται για τη συνεδρία σας καθίσει παρακαλώ. Εκείνοι που έχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις παρακαλώ σε εγκαταλείψουν την αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω ονόματι όλης της Επιτροπής. Η παρουσία σας εδώ δεν μπορώ να μην το υπογραμμίσω ότι δείχνει σε όλους μας τη σημασία που δίνουμε όλοι μας και η χώρα σας και εμείς σημασία που δίνουμε στην ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς εδώ και δύο χρόνια ήσασταν μαζί μας και σε αυτά τα δύο χρόνια συνέβησαν σημαντικά γεγονότα στη χώρα σας και, και βέβαια και στις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν οι προεδρικές εκλογές το Φεβρουάριο του 2008 και εδώ ακολούθησαν εδώ οι βουλευτές μας τον επόμενο Ιούλιο και ρίξει μια συμμαχία αν θέλετε στην που ήταν υπέρ της εισόδου της χώρας σας ε, στην Ευρώπη και στις 20 Ιουλίου ο Ράντοβαν Κάρατζης ε, μας οδήγησε σε σημαντική αλλαγή όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απαρχή της διαδικασίας και με την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και του Δικαστηρίου της Χάγης που ανέλαβε ενώματι της διεθνούς δικαιοσύνης να αποδώσει δικαιοσύνη στον αφορά τα εγκλήματα πολέμου. Ε, ξεκίνησε η δίκη και επιταχύνθηκε όμως ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διότι υπάρχει, υπάρχει κύρωση της συμφωνίας, έχει ανασταλεί η κύρωση της συμφωνίας σταθερότητας, προσωρινή συμφωνία είναι αυτή που ισχύει και την εφαρμόζει μονομερός η χώρα σας, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Οπότε έχουμε ένα κοινό συνέστημα υποστήριξης, έχουμε θετική στάση ε, έναντι μίας ε, ταχείας ε, συνάψεως αυτής της συμφωνίας. Είναι θετικός ο χαρακτήρας της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σερβία. Υιοθετήθηκε στις 14 Οκτωβρίου η έκθεση ε, υπήρξαν εξελίξεις ε, που θα θέλαμε εσάς και τους συναδέλφους σας ε, να, να παρακολουθούν αυτές τις προσπάθειες που έγιναν όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, της διαφθοράς, ε, η καταπολέμηση και μορφών υπερβολικού εθνικισμού και ρατσισμού που μπορεί να αρχίζουν να εμφανίζονται στη χώρα σας. Αυτά συμβαίνουν, αλλά θέλουμε να εκφράσουμε ε, την επιθυμία να γίνουν ακόμα μεγαλύτερε προσπάθειε σε αυτού του τομεί. Τέλο, θα ήθελα να προβώ σε μια παρατήρηση όσον αφορά σε ένα ακαθόδε θέμα ε, που ίσω να πλήττει τι ευαισθησίε κάποιων και τι δικέ ευαισθησίε, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω να το αναφέρω. Είναι το πρόβλημα του κοσυφοπεδίου. Δεν συζητούμε προφανώς την, ε, την βασική αρχή όσον αφορά το καθεστώς του κοσυφοπεδίου πλευράς Σερβίας, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει το θέμα όλους και είναι συμφέρον όλων να καταπολεμηθεί η αναρχία, να, ε, να μην υπάρχει συνεργασία μεταξύ ακραίων πολιτικών ομάδων και του οργανωμένου εγκλήματος, να μην υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης και δημόσιας ασφάλειας εκεί. Και γι' αυτό η ε, αποστολή μας της EULEX επιτόπου έχει αυτούς τους στόχους να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα, να πετύχει αυτούς τους στόχους και εντολή αυτού του φορέα μας που είναι επιτόπου θα έπρεπε και να είναι να βοηθήσει την επίτευξη των στόχων. Σκοπός της αποστολής αυτής είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, ε, να προστατευτούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στο κοσυφοπέδιο που είναι πολυεθνικό, πολυεθνωτικό μάλλον. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ και θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να σας μιλήσω σήμερα σε αυτό το σώμα που όλο και πιο σημαντικό ρόλο θα δραματίζει στην Ευρώπη της εποχής μας. Είναι μια τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητε, ε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ε, λέγοντας ότι η Σερβία είναι δεσμευμένη να εκπληρώσει την ευρωπαϊκή της ε, μοίρα, το πεπρωμένο της για λόγους γεωγραφικούς, της κληρονομιάς της, οικονομικής ευμάρειας σίγουρα, αλλά ίσως πάνω απ' όλα λόγω των ε, κοινών βασικών αξιών που πιστεύουμε ότι έχουμε. Σίγουρα οι πιο, βασικές, πιο βασικές από αυτές τις αξίες είναι να παρετηθούμε από τον πόλεμο σαν μέσο διευθέτησης διαφορών στην Ευρώπη. Πράγματι, το πρόγραμμα να, να συνδεθούν οι χώρες της, της Υπήρους αυτής ειρηνικά ε, και να σταματήσουν οι διαφορέ που έχουν χρονολογηθεί από αιώνε, οι διαρέσει και οι διαφωνίε να σταματήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τον πλούτο και την περιπλοκότητα των εθνικών παρελθόντων που ε, μα δένουν όλα αυτά σε ένα κοινό παρόν και σε ένα ε, κοινό μέλλον και πλούσιο μέλλον. Ταυτόχρονα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται τα δικαιώματα και τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν που βασίζονται στις αξίε αλληλεγγύη και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, και κοινό, ο στρατηγική, στρατηγική προτεραιότητα της Σερβίας παραμένει η πλήρης προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας για το πού πρέπει να κινηθούμε, προς τα πού πρέπει να πάμε, έχει λήξει. Δύο εθνικές εκλογές διεξήχθησαν πέρσι στη Σερβία, μία προεδρική, οι προεδρικές εκλογές και οι κοινοβουλευτικές εκλογές. Για τη χώρα μας αυτά ήταν δημοψηφίσματα, δημοψηφίσματα σχετικά με το πώς θα υπάρξει η διάδραση μεταξύ Σερβίας και του κόσμου. Οι πολίτες διάλεξαν μεταξύ δύο αντίθετων δρόμων και αποφάσισαν να ψηφίσουν υπέρ ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος. Δύο φορές το έκαναν αυτό. Η Σερβία εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, αντιμετωπίζοντας πάρα πολλά εμπόδια και καμιά φορά οι πιθανότητες ήταν επιτυχίες, ήταν πάρα πολύ μικρές. Πολλά επετέφθησαν και αυτό το δείχνει η πρόσφατη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σερβία. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά τίποτα δεν είναι τέλειο. Όμως είναι ό,τι καλύτερο είχαμε πετύχει ποτέ. Είναι, δείχνει πάρα πολύ με θετικό τρόπο τα πώς επετέφθησαν το τελευταίο δωδεκάμενο. Ενθαρρυνόμαστε πάρα πολύ από την αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρεί ότι η Σερβία είναι, έχει δεσμευτεί πλήρω ούτω ώστε να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει κάθε προσπάθεια. Υπογραμμίζοντα γενική ε, πρόοδο σε όλου του τομεί η προσωρινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι παραμένει παγωμένη και είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ικανοποιημένοι με τα συμπεράσματα τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρόσφατη δική τη διεύρυνση. Συγχαίρει τη χώρα μα, διότι εθελοντικά και παραθέτω δημιουργεί ένα ιστορικό όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων τη προσωρινή συμφωνία, ένα ιστορικό παρελθόν, και αναλαμβάνει να εφαρμόσει βασικέ πολιτικέ μεταρρυθμίσει σύμφωνα με τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Τέλο παράθεση. Θα ήθελα να τονίσω τα συμπεράσματα της στρατηγικής. Και παραθέτω, η Σερβία κατέβαλε προσπάθειες να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έχει το διοικητικό δυναμικό να σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστική πρόοδο, τέλος παράθεσης. Κυρίε και κύριοι, η Σερβία δεν έχει εστιαστεί στο να προωθήσει τις προοπτικέ της για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρώντα άλλους. Παρά τι συνεχιζόμενες δυσκολίε, επίσης προσπαθήσαμε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια να πλησιάσουν τις Βρυξέλλες και αυτό το προσπαθήσαμε μέσω τη αυξήσεω τη ε, περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε προωθήσει οικονομική ολοκλήρωση μέσω προσπάθεια δημιουργία προγραμμάτων διασυνοριακή συνεργασία όπω είναι οι διάδρομοι 7 και 10 και μέσω θεσμών όπω είναι η ΣΕΦΤΑ, η Συμφωνία για, την, ε, για το Ελεύθερο Εμπόριο στην Κεντρική Ευρώπη καθώς και η Συμφωνία για την Ενεργειακή Κοινότητα την συμφωνία για την ε, κοινότητα μεταφορών της Δυτικής Ευρώπης και η στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Δούναβη. Και η Σερβία συνέχισε να κάνει όλα ό,τι μπορούσε, ούτως ώστε η ακραία δημαγωγία να μην επηρεάζει τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων των Δυτικών Βαλκανίων. Άτομα, άνθρωποι από όλες τις πλευρές που άνθρωποι που έχουν διαπράξει φρικτά, φρικαλαία εγκλήματα πολέμου τη δεκαετία του 90 ε, και ε, δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα στην περιοχή και η Σερβία έκανε σοβαρές προσπάθειες για να καταφέρει να επιφέρει τη συμφιλίωση. Γι' αυτό ο πρόεδρος Μπόρις Τάντιτς πήγε στη Σρεμπρενίτσα στη δέκατη επέτειο ε, των ε, φοβερών εγκλημάτων πολέμου που έγιναν εκεί και υπεκλήθη στα θύματα αυτών των φρικαλαιοτήτων και γι' αυτό η Σερβία συνεργάστηκε πλήρω με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Δεν το θεωρούμε απλώ μια ε, νομική μα υποχρέωση, αλλά ηθική υποχρέωση και πολιτικό καθήκον έναντι των γειτόνων μα και του κόσμου. Αλλά πρώτιστα ε, υποχρέωση για μας, έναντι του εαυτού μας. Α μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμεί θα επιμείνουμε, θα συνεχίσουμε με το ώστε να μην ε, οι διοκόμενοι αυτοί, όσοι απομένουν και δεν έχουν συλληφθεί, να συλληφθούν. Θέλω να Στραφώ τώρα στο σημαντικότερο επίτευγμα μα αυτή τη στιγμή, η απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων διαβατηρίου. Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η Σερβία να μπει στον ε, άσπρο κατάλογο, λευκό κατάλογο Σέγγεν, έχοντα ε, εκπληρώσει ω προδιαγραφέ. Περιμένουμε μια επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο και βάσει διαβουλεύσεων βέβαια με αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν οι παρούσε προσδοκίε τελικά πραγματοποιηθούν, οι πολίτε τη Σερβία θα αρχίσουν να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Ήπειρο από 1η Πρώτου του 2010. Θα ήθελα να τονίσω ότι σχηματίζει το να μπορεί κανεί σχηματίσει μια από πρώτο χέρι εντύπωση τη Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό για του νέου τη χώρα μα που ε, αμεγάλωσαν σε μια ατμόσφαιρα πολιτική και οικονομική απομόνωση. Τώρα οι νέοι θα μπορέσουν να επισκεφθούν του ε, ε, συγγενεί του πολύ γρήγορα, να πάνε σε μια διάσκεψη στο Βερολίνο χωρί να πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να πληρώσουν το στεγαστικό του δάνειο ή να πρέπει να δείξουν το ιστορικό του τη απασχόληση για να μπορέσουν να πάνε να κολυμπήσουν στο Αιγαίο. Κυρίε και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί να ταξιδεύει κανείς ελεύθερα, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε βέβαια εκεί είναι κρίσιμη σημασία η όλη όθηση για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει αυτή η όθηση και αυτή η ορμή. Όμως φοβόμαστε ότι κάποιοι ίσως ακόμα να θεωρούν ότι ένα διάλειμμα μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση είναι μια δράση που θα πρέπει, κάτι που θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει, να κάνει ένα διάλειμμα. Καταλαβαίνω βέβαια αυτά τα συναισθήματα, όμως επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Και πιστεύω ότι τίποτα δεν θα ήταν χειρότερο από το να παγώσουμε, να κάνουμε την υπόλοιπη περιοχή να περιμένει. Ε, μια νέα ψυχολογική γραμμή διέρεσης ε, θα δημιουργεί το, το τρόπο στα Δυτικά Βαλκάνια και το κόστος όσον αφορά την αξιοπιστία της Ευρώπης ε, θα ήταν τεράστιο, απροσμέτρητο. Κόπωσης διεύρυνσης στα κράτη-μέλη θα κατέληγε σε κόπωση προσχώρησης μεταξύ των υποψηφίων εκείνων που θέλουν να προσχωρήσουν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ειλικρινά, με κάθε ειλικρινά πρέπει να πω ότι ενώ πολλοί Ευρωπαίοι μιλάνε για ε, κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις στα Βαλκάνια, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πρέπει τα Βαλκάνια να παραμείνουν το, η εκκρεμότητα της Ευρώπης. Ο ε, καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να αρχίσουμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προς, προς την πραγματική ευρωπαϊκή προσχώρηση της περιοχής. Όχι μόνο η χώρα μου να προσχωρήσει, αλλά όλη η περιοχή. Και αυτό να γίνει σύντομα, στο εγγύς μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θεωρούμε ότι έχει ανοίξει το δρόμο η Σερβή. Η Σερβία, συγγνώμη, ούτω ώστε να μπορεί να υποβάλει επίσημα την αίτησή τη η Σερβία για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό, να υποβάλουμε την αίτησή μα επίσημα μέχρι το τέλο του έτου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και καταλαβαίνουμε πώς έχουν δημιουργηθεί αυτές οι ανησυχίες. Παρ' αυτά, πιστεύουμε ότι ίγκη και είναι η ώρα να προχωρήσουμε. Κάθε κάτοικος των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κάθε προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς αυτή την κατεύθυνση και ε, με σχετική ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι, την τελευταία φορά που μίλησα στην Επιτροπή σας, σε αυτή την Επιτροπή, κάποιοι εξέφρασαν φόβους ότι η κάθετη αντίθεσή μας στο UDI, δηλαδή τη μονομερή δήλωση ανεξαρτησίας των εθνικών αλβανικών αρχών της νότιας επαρχίας του Κωσυφοπεδίου θα ήταν κάτι που θα επηρέαζε αρνητικά την περιφερειακή σταθερότητα. Αυτοί οι φόβοι δεν πραγματοποιήθηκαν. Ε, εμείς επιλέξαμε, διότι εμείς επιλέξαμε να δράσουμε υπεύθυνα. Μην αμφιβάλλετε, η βασική μας θέση όσον αφορά το κοσυφοπέδιο παραμένει ίδια. Η δημοκρατία της Σερβίας ποτέ, σε καμία περίσταση, ρητά ή ε, υπονοώντας το, θα ή έμεσα ή άμεσα θα αναγνωρίσει το UDI. Αυτή είναι η συνταγματική μας υποχρέωση καθώς και δημοκρατικό μας καθήκον. Όσον αφορά αυτό το θεμελιώδες ε, σημείο, η χώρα μας είναι ενωμένη, είναι ένα. Ταυτόχρονα υπογραμμίσαμε τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε με επικοδομητικό τρόπο, χωρίς αντιπαράθεση, μέσω διπλωματίας και μόνο στο πρόβλημα αυτό. Η απόφαση κύριε και κύριοι αποτελεί ένα αλλαγή ε, στάσης υπέρ της ειρήνης στα Βαλκάνια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχή, τη περιφέρεια αυτή, ένα θέμα με τόσο θεμελιώδη σημασία και τόσο περίπλοκα που εμπλέκει, όλους, εμπλέκει όλα τα στοιχεία, ταυτότητα, σύνορα, κοινοτικά δικαιώματα, αντίθετα ιστορικά παρελθόντα, έμεινε εκτός ε, ένοπλης ε, αντιπαράθεσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Βαλκανίων έγινε κάτι τέτοιο. Για την αρχή της σοβαρής κρίσης, ένα κομμάτι της μας ήταν να απομονώσουμε το θέμα. Για αυτό το σκοπό στραφήκαμε στα μέσα ε, ειρηνικής διευθέτησης, μέσω της ειρηνικής συνελεύσεως του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου ε, του Διεθνού Δικαστηρίου ζητήσαμε να αποφασιστεί κατά πόσο το, UDI του Κοσφοπεδίου συμφωνεί με το Διεθνέ Δίκαιο. Και μεταφέροντα αυτό το θέμα στο δικαστικό τομέα, δείξαμε πώ μπορούμε να χειριστούμε πολιτικέ διαφορέ. Κατά την άποψή μα, αυτό είναι ένα πρότυπο για επίλυση ε, σημερινών συγκρούσεων. Ένα πρότυπο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί τον κόσμο. Εκεί που υπάρχουν ε, βαθιέ διαιρέσει, όπου υπάρχει βαρύ ιστορικό παρελθόν και τα θέματα, τα προβλήματα ε, αφορούν την καρδιά του προβλήματος ε, τη εθνική ταυτότητα και καταβάλαμε σημαντικέ προσπάθειε επικοδομητικά να συνεργαστούμε με θεσμού που λειτουργούν στα πλαίσια του ψηφίσματο του Συμβουλίου Ασφαλεία 1244, όπω είναι το Γιούλεξ. Συμφωνήσαμε να εστιαστούμε στο να λύσουμε επιτόπια προβλήματα ε, ουδέτερα προ όφελο όλων των κατοίκων τη επαρχία. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία με το Ulex με επικοδομητικό τρόπο και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, πριν φτάσω στο τέλος των σχολείων μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε πρόσφατες εξε... εξελίξεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Δημοκρατία της Σερβίας θα συνεχίσει να σέβεται με ε, πλήρως ε, την ε, κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της, του γείτονά μας. Εργαζόμαστε με εκπροσώπους όλων των τριών λαών για να βρούμε μία διέξοδο ούτως ώστε να επιταχύνουμε την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της ε, ε, χώρας. Ξεκαθαρίσαμε θα υποστηρίξουμε όποια διευθέτηση είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη, τονίζοντας την ανάγκη που υπάρχει για ρεαλιστική προσέγγιση. Ε, είναι μια ευρωπαϊκή αξία του 21ου αιώνα η συνένεση, η δημιουργία συνένεσης και ε, λαμβάνεται υπόψη στις λήψεις αποφάσεων. Και θα πρέπει όλοι να συμφωνούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Καμιά φορά χρειάζεται περισσότερο χρόνο κάτι τέτοιο από ό,τι θα ήθελε κάποιο. Το έδειξε αυτό και η επικύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αλλά στο τέλο κάπου καταλήγει κανεί σε συμφωνία. Και έτσι όλοι μπορούν να προχωρήσουν μαζί. Κυρίε και κύριοι, κατά τη διάρκεια των σχολείων μου το απόγευμα ήθελα να θέσω το στρατηγικό πλαίσιο για τη μέλλον το ευρωπαϊκό της χώρας μου των Δυτικών Βαλκανίων και να τονίσω την ανάγκη να γίνουν συγκεκριμένα βήματα προς προσχώρηση. Το έκανα αυτό διότι πιστεύω ένθερμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι κάποιο που θέλει η χώρα του να προσχωρήσει, όχι γιατί φοβόμαστε να μείνουμε εκτό, αλλά από υπερηφάνεια και εμπιστοσύνη στη δυνατότητα που έχουμε να συμβάλλουμε στην πλήρη παγιοποίηση τη Ειρηνή και σταθερότητα στην γυραιά Ήπειρο. Σε μερικέ μέρε η Σερβία θα ε, συμμετάσχει στι εορτασμού για την 20η επέτειο τη πτώσεω του τείχου του Βερολίνου. Η 9η Νοεμβρίου του 1989 πάντα θα συμβολίζει αυτή την σημαντικότατη στιγμή όπου χωρίς να ακουστεί ένας πυροβολισμός έληξε ο ψυχρός πόλεμος. Για πολλούς από εμά στα Δυτικά Βαλκάνια αυτή η ημερομηνία επίσης συμβολίζει κάτι άλλο. Μια χαμένη ε, δυνατότητα, χαμένη ευκαιρία που οδήγησε σε μια μεγάλη τραγωδία. Σήμερα ο κόσμος είναι εν μέσω μιας άλλης περίοδου μεταρρυθμίσεων. Αυτή τη φορά εμείς στα Βαλκάνια είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Είμαστε αποφασισμένοι και θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Φτάνω στο τέλος των σχολείων μου και θα ήθελα να πω τα λόγια του Ζόβαν Σκέρδιτς ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς βουλευτές της Σερβίας, ο οποίος έγραψε το τέλος του περασμένου αιώνα και παραθέτω ότι να, να γίνει μια πραγματικότητα η δημοκρατία που αναπνέει θα πρέπει να ανυψώσουμε τη συνειδητοποίηση της ελευθερίας για όλους τους άντρες και γυναίκες που θέλουν να σπνεύσουν τον, τον φρέσκο αέρα της ζωής και να ζήσουν τη ζωή τους πλήρως. Για μένα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα όταν ολοκληρωθεί αυτό θα είναι θα ανυψώσει τη συνειδητοποίηση του τι είναι ελευθερία. Δηλαδή να αφήσουμε απειρχαιωμένε ιδέε όσον αφορά τη δημοκρατία σαν κάτι ουδέτερο, μια μηχανική διαδικασία. Για μένα σημαίνει να βάλουμε πιο ψηλό στόχο και να τα καταφέρουμε καλύτερα. Να θέλουμε να πετύχουμε συμφιλίωση και να οικοδομήσουμε γέφυρε. Και να βρούμε έναν τρόπο να ζήσουμε τη ζωή μα αλληλέγγυα ο ένα με τον άλλον μέσα σε μια κοινωνία κοινών αξιών που είναι ψηλέ και βαθιέ σημαντικές αξίες και κοινά συμφέροντα που, που είναι δίκες και μας εμπνέουν αυτές οι αξίες. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Και έχω κάθε πεποίθηση ότι θα αρπάξουμε αυτή τη στατηγική ευκαιρία που προσφέρεται στους γενναίους. Είναι η ώρα μας να αρπάξουμε την ευκαιρία και να την θρέψουμε και να την τροφοδοτήσουμε ώστε να δυναμώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πραγματικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και ξεκινάμε τη συζήτηση. Δίνω το λόγο πρώτης στον εισηγητή κύριο Κάτσιν παρακαλώντας να παραμείνει στο χρονικό όριο του τριλέπτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρία πρέσβία, θα ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ για τα όσα μπορέσατε ήδη να επιτύχετε για, στα, στα πλαίσια του οδικού χάρτη ήδη η Σερβία κατάργηση της προξενικής θεωρήσεις. Τώρα το πότε θα απολαύσουν τα ωφέλη αυτά οι πολίτες είναι θέμα προθεσμίας, είναι θέμα ημερομηνία. Θα χαρώ πάρα πολύ να, έλθουν, να μπορούν να έλθουν ε, να μας επισκεφθούν οι Σέρβοι πολίτες χωρίς προξενικές θεωρήσεις. Νομίζω ότι δουλέψατε καλά και αποδείχνετε ότι η Σερβία έλαβε μια όταν παίρνει μια απόφαση μπορεί πράγματι και την υλοποιεί. Σας συγχαίρω επίσης και για το ότι η Βοηβοδίνα επιτέλου αποκτά καθεστώ. Και ήδη η Σερβία προχωρεί με ταχαία βήματα. Χρειάζεται νέες περιφέρειες η ε, Σερβία και οι περιφέρειες αυτές χρειάζονται υποστήριξη για να εξασφαλίσουν συνοχή και συνεργασία. Η Σερβία πρέπει να είναι κράτος δικαίου. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση για όλους. Ο ποινικό κώδικας της Σερβικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να παραβιάζεται από κανένα. Γι' αυτό και <clears throat> επισημαίνω ορισμένες ε, περιπτώσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων που ε, διαμηνύουν κάποιες ε, μη κρατικέ οργανώσεις μια κυρίαρχη χώρα ελέγχει το εδαφός της και είμαι βέβαιος ότι το πράττει η Σερβική Δημοκρατία, ότι έχει τον έλεγχο δηλαδή σε ολόκληρη την επικράτειά της. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί τελικά ο Μλάντιτς και θα καταλήξει ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Χαίρομαι που η Σερβία συνεργάζεται όχι μόνο με το Δικαστήριο της Χάγης αλλά και με άλλες χώρες όπως τη Σλοβενία. Η Σερβία είναι η μεγαλύτερη χώρα της ε, περιοχής αυτής και επειδή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη χώρα έχει και σημαντικό ρόλο να παίξει ανάλογο, ε, τηρωμένο των αναλογιών βεβαίως, του ρόλου που μπορεί να παίξει, που παίζει η Γερμανία και η Γαλλία στην ε, Ενωμένη Ευρώπη. Η πρόοδος η δική σας θα ωφελήσει και τους υπόλοιπους γειτονές σας ενώ οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση θα ε, τους βλάψει. Γι' αυτό και χαίρομαι για την ε, συμφωνία σας με την ε, Ιούλεξ που αποτελεί σημαντική πρόοδο για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος και στο Κόσοβο. Εξάλλου, ως εισηγητής θα σας πω ότι εμείς αναμένουμε από τη σερβική κυβέρνηση να ζητήσει από, το σερβικό πληθυσμό του Κωσόβου να συμμετάσχει στις εκλογές. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις ε, περιφερειακές αυτές εκλογές και να συμμετάσχουν στο πολιτικό γίγνεσθε. Εν τέλει, το εξή, κύριε ε, Υπουργέ. Όπως είπατε, το μέλλον ανήκει στους θαραλέους. Είμαι ε, βέβαιος ότι υπάρχει πολιτικό θάρρος στη Σερβία ώστε να ξεκινήσουν βήματα τα οποία θα μας εκπλήξουν θετικά και τα οποία θα μας πείσουν ότι ο φόβος ότι η, ο φόβος που λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν θα διευρυνθεί πέραν της Κροατίας είναι ε, ψευδής. Η Σερβία δεν μπορεί να αποτελέσει όμοιρο της ιστορίας της. Δείξτε μας λοιπόν με τις προσπάθειες που θα καταβάλλετε ότι το μέλλον σας βρίσκεται στην Ευρώπη, όπως το μέλλον, το, το μέλλον των Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κάτσιν. Ο πρόεδρος Υποπιτροπής Άμυνας Ντανζά έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Δεν ακούγεται τίποτα πριν. Σας ε, ευχαριστούμε για αυτά που είπατε και για την ε, πεποίθηση και σας και της κυβέρνησής της ότι θα πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα για να μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία. Η κυβέρνησή σας, πρέπει να πω, εξελέγει όπως και ο πρόεδρος Τάντιτς το 2008 βάσει ενός προγράμματος χωρίς αμφισημίες με απόλυτη προτεραιότητα προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θυμούμε ότι τότε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θεωρήθηκαν από κάποιους ως δημοψήφισμα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από άλλους, από άλλα θέματα. Και αυτοί που πρέσβευαν το αντίθετο από εσά δεν κέρδισαν. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω λοιπόν για αυτή την πλευρά που τονίζει θετική όσον αφορά την, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να πω ότι κατασπαταλάτε πολύ μεγάλη διπλωματική ενέργεια για το θέμα του κοσυφοπεδίου. Είπατε ότι θα θέλετε να μιλήσετε μόνο από νομικής σκοπιάς μετά από κάποιες δράσεις και διακηρύξεις της κυβέρνησης της Σερβίας. Επιτρέψτε να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες. Και φαίνεται ότι συγχρόνως με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλετε να δώσετε και προτεραιότητα στο θέμα του κοσυφοπεδίου. Πρέπει να σας πω ότι 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου και δεν θα υπαναχωρήσουν. Πώς μπορείτε λοιπόν να διαχειριστείτε αυτή την ε, ένταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο προτεραιοτήτων. Επίσης, αναφέρατε στα πλαίσια της ε, διεύρυνσης και τώρα μιλώ εξ ονόματος ε, του κόμματός μου, του Προέδρου Σαρκοζή, ότι για μας δεν υπάρχει αμφισημία στρατηγική και πολιτική για οποιαδήποτε χώρα της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της ε, Σερβίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Νταουζά. Ο κύριος Τάλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρέσβερα, καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ, στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι πολύ σημαντική. Γίνεται προσπάθεια να προωθήσουμε την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε και συζητήσαμε σήμερα την έκθεση για την πρόοδο τη Κροατία. Και κλείνουμε τώρα και επίση τη πρώην ε, Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Ε, ε, κλείνουμε τώρα τον κύκλο αυτόν με την δική σας χώρα. Και τη ευχόμαστε να μπορέσει να ενταχθεί. Ε, έχω μια ερώτηση. Γνωρίζουμε ποιο είναι ο ουσιαστικό και ποιο είναι ο τυπικός λόγος για την μη εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και συνεργασίας με την ε, Σερβία. Δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η Σερβία πραγματικά αναζητεί και ψάχνει να βρει τον Βλάντιτς και τον Χάτσιτς. Είναι, είναι απαραίτητο να εκπληρώσει αυτή την, αυτή την υποχρέωση. Πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. Από τον κύριο Τρόγνιακ ακούσαμε χθε ότι η Κροατία και η Σερβία το Ζάγκρε πρότεινε δηλαδή στο Βελιγράδι να συμφωνήσουν πάνω σε μια οριακή γραμμή όπου το μεγαλύτερο μέρος της θα περνάει από το Δούναβι ανάμεσα στις δύο χώρες. Εκεί υπάρχουν ε, παραδοσιακά προβλήματα σε σχέση με το κτηματολόγιο και άλλα. Πού βρίσκεστε με το θέμα αυτό. Είστε διατεθειμένοι να το επιλύστε το δυνατόν συντομότερο ώστε να μην αποβεί ένα κόλλημα για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Δανά. Η κυρία Κύριε Υπουργέ, για πρώτη φορά σας γνωρίζω, είμαι νέη εισηγήτρια για το Κόσοβο. Στο σύντομο αυτό δίλεπτο θα ε, ρίξω το βάρος μου σε αυτό το ε, θέμα. Είπατε και ε, πραγματικά με εκπλήξατε με τα θαυμάσια αγγλικά σας και με τη θαυμάσια ρητορική σας ικανότητα. Είπατε ότι ο πόλεμος τέλειωσε. Μιλάμε για ειρήνη, για σταθερότητα. Και εγώ το πιστεύω αυτό και ξέρω ότι το πιστεύει και ο πρόεδρος σας. Συμφωνούμε λοιπόν εδώ. Όταν λέτε ότι η χώρα σας είναι ενωμένη ε, επί του θέματος της μονομερούς δήλωσης ανεξαρτησίας του Κωσόβου, ξέρω ότι και στην χώρα σας που υποστήριξε τους ε, Σέρβους κοσοβάρους να χρησιμοποιήσουν τις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου για να πάρουν τα πράγματα, τα τοπικά πράγματα στα χέρια τους. Θα ήθελα να σας ζητήσω από τους Σέρβους κοσοβάρους να ζητήσετε κι εσείς να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει την αποκέντρωση τους πολίτες, τους Σέρβους Κωσοβάρους, τους πολίτες αυτής της χώρας να μπορέσουν να ε, πάρουν στα χέρια τους τις πολιτικές στο τοπικό επίπεδο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι οι πολίτες σας θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Εγώ αγωνίστηκα υπέρ αυτή τη δυνατότητα και στην Εθνική μου Βουλή για 10 χρόνια που ήμουν βουλευτή τη Αυστριακή Βουλή. Όμω υπάρχουν οι συνολικοί ελέγχοι και προ το Κόσοβο θα παραμείνουν οι ελέγχοι αυτοί όπως σε κάθε διεθνές ε, σύνορο. Και αυτό είναι σημαντικό. Τέλος, τι γίνεται με την κατάσταση στην Μητροβίτσα. Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα που έχετε να πιέσετε και την ευρωπαϊκή σας προοπτική για να διευκολύνετε την ένταξη και των ανθρώπων στην περιοχή αυτή. Ξέρω ότι είπατε ότι η ε, Σερβία ποτέ ρητά ή σιωπηρά δεν θα αναγνωρίσει την μονομερή δήλωση. Ίσως στην πολιτική το να λέει κανείς ποτέ δεν είναι τόσο σωστό όταν εξετάζει ένα κοινό μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Τάνοκ. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών σε μια θαυμάσια, γλω... σε μια θαυμάσια παρουσία σας στην στην γλώσσα του Σέξπιρ ή μάλλον στη βορειοαμερικανική εκδοχή της γλώσσας του Σέξπιρ. Εγώ είμαι ένθερμος οπαδός της χώρας σας και ε, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να ξεφύγετε από τις συνέπειες ε, των πολέμων και του ακραίου εθνικισμού. Ε, με ανισχύει και μένα η κατάσταση προέκυψε μετά από την μονομερή δήλωση ανεξαρτησίας ε, του Κωσόβου, επίση με τις εξελίξεις στο Νότιο Κάφκασο και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά ε, σημαίνουν σημαντικά προβλήματα και για το μέλλον και για την περιφερειακή σταθερότητα. Προσωπικά, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη και όχι του κόμματος μου είτε της πολιτικής μου ομάδας, της ECR, Πιστεύω ότι ε, το θέμα του Κωσόβου έπρεπε να είχε διαρευνηθεί περισσότερο. Έχουμε τώρα μια de facto κατάσταση στην Πιτροπίτσα που δεν μπορεί να επιληθεί με ικανοποιητικό τρόπο. Έχουμε μείνει λοιπόν με την ε, δύσκολη αυτή κατάσταση στα χέρια μας. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο για το προσεχές μέλλον. Εγώ είμαι εισηγητής για το Μαυροβούνιο που ο Όλι πρόσφατα εδώ στην παρούσα επιτροπή είπε ότι είναι Καλά τα νέα, διότι προχωρεί καλά προ την κατεύθυνση να ενταχθεί. Θα ήθελα να ακούσω, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, για τι διμερείς σχέσει μεταξύ Σερβία και Μαυροβουνίου και κατά πόσον μπορείτε εσεί να συντονίσετε τις ε, διαπραγματεύσει όταν θα λάβετε το καθεστώ της υποψήφια χώρας και τις επικαλύψεις που υπάρχουν με την πορεία του Μαυροβουνίου. Η Μαυροβουνίου είναι μικρή χώρα με περιορισμένους πόρους Αναγνωρίζω ότι κάθε χώρα βεβαίω πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με τα όσα επιτυγχάνει η ίδια για την πλήρωση των κριτήρων τη Κοπενχάγη. Αλλά κατά πόσο μπορείτε να συνδυαστείτε, πόσο μπορεί να υπάρξει συνδυασμό των προσπαθειών μεταξύ Ποντγκόριτσα και Βελιγραδίου. Ευχαριστώ κύριε Τάνο. Ο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ε, μάλλον Αγκουράκη είπατε κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Ναι, μάλλον κύριο Αγκουράκη εννοούσε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θέλω και εγώ να χαιρετήσω τον ε, Υπουργό και την ε, πρέσβυρα ε, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, να τους μεταφέρω τους χαιρετισμού και τις καλύτερε ευχές των Ελλήνων. Θα μου επιτρέψουν δύο-τρία σχόλια ο κύριος Υπουργό στην παρέμβασή του. Το πρώτο είναι ευπρόζεκτη φίλη μας από τη Σερβία, όχι μόνο για μπάνιο στο Αιγαίο όπως είπε στην Ελλάδα, ε, ελπίζω με τις διευθετήσεις που θα υπάρχουν να έρχονται και πιο συχνά και να παραμένουν και περισσότερο χρονικό διάστημα γιατί φαντάζομαι θα το θέλουν και για οικονομικούς λόγους με δεδομένο ότι η κατάσταση στη χώρα τους δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη όπως και στην Ελλάδα εξάλλου και ίσως ο κύριος ε, Υπουργό να μπορέσει να δώσει και κάποιες εξηγήσει οικονομικά προς τα που θα πάει η Σερβία και πώς. Αυτό ήταν ένα πρώτο θέμα που ήθελα να θίξω. Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να τον ρωτήσω και το σχόλιο του είναι ότι με την, ε, ε φέτος συμπληρώνονται και 10 χρόνια από τους νατοικούς βομβαρδισμούς ε, στη Ιουγκοσλαβία. Από αυτόν τον ε, φοβερό πόλεμο, τον απαράδεκτο που έγινε εκ μέρους του ΝΑΤΟ και ο οποίος βεβαίως οδήγησε και σε μια τραγική κατάσταση και στη χώρα του αλλά συνολικά στα Βαλκάνια. Το οποίο αποτέλεσμα ήταν και η απόσχεση του Κωσόβου. Άρα το θέμα της αλλαγής συνόρων δεν είναι ότι λύνεται στην Ευρώπη χωρίς πολέμους και αιματοχυσία. Και χαίρομαι για τη δήλωση που έχει κάνει ότι η Σερβία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει την απόσχηση του Κωσόβου γιατί πρόκειται για μια παράνομη πράξη και έκθεση εξάλλου το τεκμηριώνει αυτό κατά τη γνώμη μα. Αλλά το ερώτημα είναι τι θα κάνει για να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα ευχαρίστως. Υποστηρίζω και την πολιτική σας δέσμευση για μια ενταξιακή πορεία. Στα ωραία αμερικάνικα αγγλικά σας μας είπατε ακριβώς όλα όσα θα θέλαμε να ακούσουμε. Συμφωνώ επίσης ότι οι άνθρωποι στην ε, Σερβία σε μεγάλη πλειοψηφία θέλουν μια πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή και διότι έχουν παραπλανηθεί κατά επανάληψη από τι ηγεσίες του στο παρελθόν και στην κατεύθυνσή του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω ότι τέτοιε παραπλανήσεις δεν θα επαναληφθούν. Ελπίζω άλλωστε υπέρ των Σέρβων να μπορούν πράγματι σύντομα να ε, ε, διακινούνται ελεύθερα. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ακόμα ορισμένα χρόνια σε σχέση δηλαδή με το Κόσοβο για να αναγνωρίσετε την πραγματικότητα. Είπε και η κυρία Λούνατσεκ, μην λέτε ποτέ, ποτέ στην πολιτική και ιδίω στα Βαλκάνια. Πάντως, πριν από τις κοινοτικές εκλογές στο Κόσοβο, ξαναθέτω το ερώτημα, μπορούμε να αναμένουμε από εσάς επισήμως προτροπή προς τους Σέρβους Κοσοβάρους να συμμετάσχουν στις κοινοτικές εκλογές, στις δημοτικές, τοπικές εκλογές, δηλαδή στο Κόσοβο, εάν δεν συμβεί αυτό ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουν οι Σέρβοι Κωσοβάροι αν δεν συμμετάσχουν στις ε, κοινοτικέ εκλογές εκεί, κατά την άποψή σα. Και τέλος, για Μλάντιτς και Χάτσιτς. Νομίζω ότι γνωρίζετε, ότι εμείς γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν αρκετές και επαρκείς δομέ στην Σερβία που προστατεύουν τους Μλάντιτς, Χάτσιτς και διαφορου άλλου ενώ γνωρίζουν πού ακριβώ βρίσκονται. Και το ερώτημα είναι, έχετε πολιτικά φόβο να τους συλλάβετε και να τους παραδώσετε ή φοβάστε ότι ενδεχομένως κινδυνεύετε και εσείς οι ίδιοι γιατί και παλαιότερα έχουν δολοφονηθεί ε, οι ηγέτες σας. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Με σας κλείνει ο πρώτος γύρος παρεμβάσεων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό και μετά θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια. Όντως είδατε ότι υπάρχει πρόοδο στη Σερβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τον κύριο Κατσίν που το επιστώνει και είμαστε. Να συνεργαστούμε και να γίνουμε και με όλους τους βουλευτές ώστε να μπορέσει να διευκολυνθεί η προσχώρηση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω αυτό το πάγωμα. Όντως έχει παγώσει όλη η διαδικασία. Και τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τη συνεργασία με τη Χάγη. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο είπα προηγουμένως. Πλήρως και χωρίς αμφισημίες έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις ώστε να μην υπάρχουν ε, ένοχοι οι οποίοι θα αποφύγουν τη δικαιοσύνη. 44 από 46 έχουν προσαχθεί στη ισογενική κυβέρνηση. Η Σερβία κάνει ό,τι μπορεί και παρέδωσε και τον Κάρατζιτς. Και αν αυτό δεν συνέβη, όπως λέτε, για πολιτικ... είχαμε πολιτικούς φόβους, δεν έχει Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο από αυτό το οποίο κάνουμε τώρα για να εξασφαλίσουμε ότι θα ευρεθούν οι ένοχοι, θα συλληφθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους σε ένα κανονικό δικαστήριο. Και όπως είπα στην εισαγωγή μου, δεν θα σταματήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν άτομα στην Σερβία που υποστηρίζουν τη θέση της κυβέρνησης. Υπάρχουν άλλοι που μας μισούν εξαιτίας αυτής της θέσης. Όλοι όμως, όσοι μας υποστηρίζουν ή μας μισούν, είναι ενωμένοι, διότι ξέρουν ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γίνει και σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι σε αφορά την προσπάθεια. Όπως σας είπα, όλο και λιγότεροι συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Εισαγγελέα του κυρίου Μπράμοβ έχουν ε, εκφράζουν αμφιβολίες ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και από πολιτική σκοπιά και από πρακτική. Ο κύριος Μπράμιτς αυτή τη στιγμή είναι στο Βελιγράδι. Ενημερώθηκε για την όλη κατάσταση από τις δικές μας υπηρεσίες και σύντομα θα υποβάλει νέα έκθεση. Ελπίζω ότι η έκθεση θα αντικατοπτρίζει τη θέση μας. Ακόμη και την τελευταία φορά που υπήρχε δυνατότητα από τον κύριο Μπράμιτς να ενημερώσει τους υπέξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τέτοια ερώτηση αν πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση που δεν το κάνει τώρα απήντησε αρνητικά. Ελπίζω λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή δεν θα διανυστεί. Κατανοώ κάποιες ευαισθησίες Όντως τις κατανοώ. Όλοι είμαστε πολιτικοί και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πολιτική με ήττα στις χώρες μας. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής και να το σκεφτείτε. Η Κροατία βρίσκεται στον καλύτερο δυνατό δρόμο να προσχωρήσει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα. Για μας, για τη Σερβία, για την Ευρώπη και βεβαίως για την περιοχή. Μετά λοιπόν από την προσχώρηση της Κροατίας θα πω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία πάυση. Πολλοί το πιστεύουν αυτό και το λένε. Και υπάρχει μία λογική που άπτεται και αυτού του επιχειρήματος. Υπάρχει ανάγκη παύσης μετά την Κροατία. Αν μπορέσετε να συνδυάσετε το μήνυμα αυτό με την πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας Φανταστείτε πώς εμείς σκεφτόμαστε στα Δυτικά Βαλκάνια που είμαστε εδώ και 500 χρόνια στο ίδιο πλοίο με την Τουρκία. Πιστεύουν κάποιοι ότι και τώρα θέλουμε να μπούμε στο ίδιο πλοίο. Και βεβαίω κάποιοι που πέρασαν την περισσότερη ζωή του σε μια τέτοια κατάσταση έχουν αυτή την άποψη, αλλά δεν είναι έτσι. Μην κάνετε και εμά να περιμένουμε τόσα πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μετά αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε δύσκολα τα πράγματα, αλλά θέλουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, διότι πιστεύουμε ακόμα κράδαντα στην πλήρη συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής και όσον αφορά τους εγκληματίες πολέμου θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να έχουν το δικαίωμα εκεί να εξηγήσουν γιατί το έκαναν αυτό. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν για το Κωσυφοπαίδιο και προφανώς θα πρέπει να καταναλώσω χρόνο για να τα απαντήσω. Πολλοί είπαν ότι η Σερβία είναι η χώρα κλειδί όσον αφορά τη στρατηγική ε, στην περιοχή. Και αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονό ότι έχουμε δύο εισηγητέ για αυτό το θέμα. Τον κύριο Κατσίν και την κυρία Λούνατσεκ. Έτσι το εκλαμβάνουμε εμείς το γεγονό ότι υπάρχουν δύο εισηγητές. Θα συνεργαστούμε και με τους δυο σας. Όντως. Λαμβάνουμε την κατάσταση του κοσυφοπεδίου πάρα πολύ σοβαρά και θέλω και πάλι να επαναλάβω ότι, ότι μετά από αυτή την μονομερή ε, δήλωση δια... Ε, ανεξαρτησίας θα υπήρχαν πολλά προβλήματα και διαμάχες. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, αποφάσισε η Σερβία ότι αρκούν οι φιλονικίες, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδό και είπαμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διεθνείς ε, όλα τα διεθνή θεσμικά όργανα, όλους τους οργανισμούς, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Πάρα πολύ λίγοι στον κόσμο μπορούν να πούν κάτι κατά του δικαιώματος μιας χώρας να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο και να δούμε πώς θα γνωμοδοτήσει το αυτού του θέματος. Τι θα κάνετε θα μου πείτε αν πει η απόφαση αυτή ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σωστά έγινε αυτή η μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας. Θα το ακολουθήσουμε. Αν μας πούνε ότι πρόκειται για παραβίαση, θα το ακολουθήσουμε επίσης. Θα ασκήσουμε όμως ως κυρίαρχη χώρα αυτό το, δικο, το κυρίαρχο δικαίωμά μας να, να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και την εδαφική μας ακαιρεότητα. Στο Κωσυφοπέδιο ή όπου και να ζει κάποιος, στην υπόλοιπη περιοχή, υπόλοιπες περιοχές γειτονικές, στην Σερβία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την μπορούμε να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Όταν ληφθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Και να λέγεται ότι ποτέ δεν πρέπει κανείς να λέει ποτέ συμφωνώ. Αλλά είσαι όλα είσαι τίποτα. Όχι μόνο για την αναγνώριση του κοσυφοπεδίου από την Σερβία, για οτιδήποτε συμβαίνει. Τι είναι λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να προωθήσουμε την ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής, να προσχωρήσουν αν θέλουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής και πιστεύω ότι και το κλίμα που θα διαμορφωθεί θα είναι όλο και περισσότερο κλίμα θετικό και κλίμα εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω ποιες λύσεις θα ακολουθηθούν, αλλά πιστεύω ότι κάποια συμβασμός θα μπορέσει ίσως να εξευρεθεί στο μέλλον. Όντως, επενδύουμε πολλά στις διπλωματικές ενέργειες που ε, αναλαμβάνουμε για το κοσυφοπαίδιο. Νομίζω ότι και εκείνοι ως χώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν για να ε, μπορέσουν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία και μας. Όσο λοιπόν εξασφαλίζεται ένα κλίμα ειρήνης και ανέμακτος πορεία νομίζω ότι θα πάμε καλά. Και βεβαίως εκτιμώ το ότι η διαδικασία προσχώρησης της Σερβίας όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι διαφορετικό από το θέμα του κοσυφοπεδίου και του καθεστώτος της χώρας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο όσο προχωρούμε, όπως είπα, τα πράγματα ελπίζω ότι όλο και περισσότερο θα βελτιώνονται. Δεν ήταν πλώς και μόνο δυνατόν για τη Σερβία να μπορέσει να συμφωνήσει με τις τοπικές εκλογές οι οποίες έγιναν οι οποίες ε, αναγγέλθηκαν πριν από μερικούς μήνες και θα γίνουν στο Κωσυφοπέδιο στις 15 Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ κακή ιδέα να αναγγελθούν εκλογές εκτός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 444. Έπρεπε να γίνουν τα πράγματα χωρίς να παραβιαστούν οι αποφάσεις του σχετικού ψηφίσματος σχετικής απόφασης των Εθνών. Δεν ήταν δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, απλώς δεν συνέβη. Δεν μπορεί λοιπόν κάτι τέτοιο να το εγκρίνει η κυβέρνηση της Σερβίας, διότι κάτι τέτοιο σε παραβίωση της απόφασης των ΗΠΑ για το 1244 και όχι στο πλαίσιο αυτής της ε, ε, απόφασης και σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοσφοπεδίου είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν με ευχαριστεί αυτή η κατάσταση και να πρέπει να σας αναλύσω αυτή τη θέση της Σερβίας. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν μπορούσε να βρεθεί μια άλλη λύση για να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Πριν από τέσσερα χρόνια, ο πρόεδρος της Σερβίας ενέκρινε τη διενέργεια τοπικών εκλογών. Ήταν ανεπιτυχές το Όλαγχη. Την τελευταία φορά που υποστηρίξαμε κάτι τέτοιο, μόνο πολύ λίγοι Σέρβοι ε, συμμετείχαν. Ίσως το 0,5% της ε, Έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο τώρα είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα επιθυμούσα να γίνουν τα πράγματα με διαφορετικές συνθήκες. Τώρα, μιλώντας για αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ αυτών των εκλογών Σερβία, γιατί κάποιος το ανέφερε και κάποιοι όντως υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχε Αλβανού στην κυβέρνησή του ο Μιλόσεβιτς. Και στη δεκαετία του 90 και εκείνοι συμφωνούσαν την πολιτική του νόμου του Μιλόσεβιτς. δεν ανταποκρίνονταν ίσως όμως στην πλειοψηφία των επιθυμιών των δικών τους. Η δημοκρατική νομιμότητα είναι κάτι το σημαντικό και στην συγκεκριμένη περίπτωση ελείπει. Πρόκειται λοιπόν για μια δύσκολη κατάσταση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να την ξεπεράσουμε. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον μετά την διενέργεια αυτών των εκλογών Θα αρχίσουμε διάλογο που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε επίλυση των προβλημάτων με την εκπροσώπηση ατόμων της τομικών κοινιών που δεν θα καταπατά και δεν θα παροφιάζει το δίκαιο και τους νόμους. Εμείς συνεχίζω να λέω ότι θέλουμε να συναντούμε τη διεθνή κοινότητα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να ομαλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο δεύτερος γύρος παρεμβάσεων δυστυχώς θα πρέπει να μειωθεί στο 1,5 λεπτό για καθέναν. Αν θέλουμε να προσθεθούν και άλλοι συνάδελφοι και αν θέλουμε να τηρήσουμε το ωράριο. 1,5 λεπτό λοιπόν. Ο κύριος Τκάνοκ, δεν απαντήσατε για το Μαυροβούνιο και τις σχέσεις με τη Σερβία. Συγγνώμη, λέει ο υπουργό. Ναι, ναι, ναι, παρασύρθηκα, συγγνώμη. Και το Κωσυφοπέδιο. Ναι, συγγνώμη, λέει ο υπουργό. Ε, κοιτάξτε. Ο πρεσβευτής του Μαυροβουνίου χτες παρουσίασε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρό μας και νομίζω ότι περνάμε μια φάση σχέσεων Μαυροβουνίου-Σερβίας που είναι μια φάση ανάκαμψης των σχέσεων αφού χάσαμε πολύ εμπιστοσύνη αφού η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου πέρσι αποφάσισε να αναγνωρίσει τη μονομερή ε, διακήρυξη ε, ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. Μία μέρα μετά την ε, ψηφοφορία στην στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που μεταβίβασε το θέμα στο δικαστήριο και θεωρήσαμε εμεί ότι ήταν πολύ κακός ο χρονισμό αυτός. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Επί αιώνε έχει κρατήσει αυτή η σχέση. Οι αναγνωρίσεις του Κωσυφοπεδίου από το Μαυροβούνιο ε, δεν ήταν μια απλή αναγνώριση για τη Σερβία. Να το πω ειλικρινά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με έναν τρόπο που δεν είναι εις βάρος της ιδιαίτερης ειδική αυτής σχέσης. Όσον αφορά την παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη, όλα αυτά τα ζητήματα, η πολιτική της Σερβίας προς το Μαυροβούνιο δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Μαυροβούνιο, διότι πάντα το Μαυροβούνιο θα είναι η εγκύτερη χώρα, κράτος, έθνος, όπως θέλετε. Έτσι ήταν επί αιώνες. και δεν αναμένεται να αλλάξει. Υπάρχουν οι πολιτικές διαφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση που επικρατεί στο Μαυροβούνιο για τους ε, ε, Σέρβους που ζουν εκεί και Ελπίζουμε ότι με κοινέ προσπάθειες με την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου θα βελτιωθεί η κατάσταση. Όσον αφορά τις προοπτικές του Μαυροβουνίου για προσχώρηση στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι κάνουμε θα τους το διαθέσουμε. Ε, ε, θα, θα είναι πιο εύκολα τα μεταφραστικά ζητήματα, διότι μιλάμε την ίδια ή πολύ παρόμοια θα έλεγαν ε, κάποιοι, γλώσσα. Οπότε θα βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο όσο μπορούμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι είναι γείτονέ μας. Δεν έχουμε πιο κοντινό και σημαντικό γείτονα από το Μαυροβούνιο ανταγωνίζονται τη Βοσνία στον αφορά αυτό. Και η Βοσνία και το Μαυροβούνιο είναι σημαντικότατοι καλοί γείτονε, με του οποίου γείτονε θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τι καλύτερε δυνατέ σχέσει. Ό,τι και να συμβεί. κυρία Ντεκάιζερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους συγχαίροντάς σας για την πρόοδο που επιτέχθηκε στη χώρα σας, για την προσχώρησή σας στην Ευρώπη και τον εκδημοκρατισμό. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Μα σαν ανησυχεί η κατάσταση για τον Μπλάντιξ, και τον Χάτζιτ, που δεν έχουν ακόμη συλληφθεί. Και είπατε εσείς πλέον τις μιας φορές ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι στα χέρια μας. Τι δεν είναι στα χέρια σας. Τι δεν μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή ποια είναι τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζετε. Δεύτερο ερώτημα, πάρα πολύ οδυνηρό. Η δίκη του Κάρατζιτς μέσω μαρτυριών μας θυμίζει άσχημες καταστάσεις και όπως ξέρετε εμείς έχουμε κάνει και μία σε σχέση με την Σρεμπενίτσα και την κατάσταση που είναι εκεί. Γιατί ποτέ λοιπόν το δικό σας κοινοβούλιο για την γενοκτονία στη Σρεμπένιτσα δεν έχετε υιοθετήσει ψήφισμα και δεν έχετε ποτέ καταδικάσει την ε, στάση του σερβικού στρατού προς τους μουσουλμάνους. Νομίζω ότι για να μπορέσει να υπάρχει κάποιος, ε, ε, κάποια ανακούφιση, κάποιος εφησυχασμός δεδομένου ότι είναι πολύ νοπά τα αποτελέσματα της κατάστασης στις μνήμες, γιατί δεν κάνετε κάτι. Επίσης, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με το κοσυφοπαίδιο, το οποίο λέγει ότι εκείνο προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα προς τη δική σας κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάιζερ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Λάτφορντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Θα συγχαρώ τη Σερβία για την επιτευχθήσα πρόοδο. Ευπρόσδεκτα αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών. Λέτε ότι δεν υποστηρίζει το, την προσχώρηση της Σερβίας βάρος άλλων και ότι η προσχώρηση της Βοσνίας Εζεγοβίνης ήταν στατηγική προτεραιότητα για σας. Στα πλαίσια της απελευθερώσεως των προξενικών θεωρήσεων, κάτι που υποστηρίζει το Κοινοβούλιο και για τα πέντε κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, θεώρησα λίγο ότι τα μαυρώσατε αυτό, αυτό που είπατε μετά ότι η πρεσβεία σας εδώ στις Βρυξέλλες πίεζε τους ευρωβουλευτές κατά της προσέγγισης που ακολουθούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να ε, υποστηριχθεί η απελευθέρωση θεωρήσεων για τις χώρες συμπεριλαμβανομένης τη Σερβίας και εντός του πεδίου εφαρμογή να μπει η Αλβανία και η Βοσνία Ζεγοβίνη. Εσείς επιμένατε ότι δεν θα πρέπει να απελευθερωθεί η θεώρηση μάλλον εμείς λέγαμε ότι πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια αυτές οι χώρες για να απελευθερωθεί το καθεστώς θεωρήσεων. Η πρεσβεία σας πίεζε τους ευρωβουλευτές κατά της προσέγγισης μας να διευκολύνουμε αυτές τις δύο χώρες. Συμφωνώ με την κυρία Τεκάιζερ. Δεν καταλαβαίνω όταν κάνετε ό,τι μπορείτε. Η χώρα σας ακόμα δεν βρίσκει αυτούς που διώκονται και πώς η Σερβία ε, στον οδικό χάρτη τον των θεωρήσεων ε, συμμορφώθηκε όσον αφορά τις προδιαγραφές που υπάρχουν για την ασφάλεια, δικαιοσύνη κλπ. όταν δεν μπορείτε να συλλάβετε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ κυρία Λούτφορ. Πρέντα για μισή λεπτό κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, <clears throat> ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι που η έκθεση πρόοδου της Σερβίας είναι τόσο θετική. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τις σχετικές συμφωνίες το δυνατόν συντομότερο, ώστε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της σερβικής κυβέρνησης. Νομίζω επίσης ότι ήταν σημαντικό που δόθηκαν οι ελαφρύνσεις για τις ε, προξενικές θεωρήσεις, για, το σύστημα Visa δηλαδή, γιατί διευκολύνουν τους πολίτες να διακινούνται και να έρχονται και στην Ευρώπη. Έχω μια ερώτηση προς τον Υπουργό. Από τον Οκτώβριο λέμε ότι η σερβική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την προστασία των μειονοτήτων. Υπάρχουν όμως ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τις δραστηριότητες της κυβέρνησης απέναντι στη ρουμανική μειονότητα. Τι προτίθεται να κάνει η σερβική κυβέρνηση ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση της ρουμανικής μειονότητας στην Σερβία. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κοπά έχει το λόγο. Ε, θέλω και εγώ να καλωσορίσω εκ μέρους του, της πολιτικής μου ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τον Υπουργό και να χαιρετήσουμε τα σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει από τη χώρα τους. Νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέει ο Υπουργό ότι η Σερβία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα διάλογο με το Κόσοβο. Πρώτη ερώτηση, αν αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνει πριν την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Δεύτερο σημείο είναι σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο κύριος Μπράμερτς στην προηγούμενη του έκθεση σημείωσε την σημαντική πρόοδο. Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας επίσης μιλάει για τις προσπάθειες Σερβίας να εντοπίσει και να παραπέμψει ε, στη δικαιοσύνη τους τελευταίους εγκληματίες πολέμου που έχει μείνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η κυβέρνηση έχει κάτι συγκεκριμένο να παρουσιάσει στον ειδικό εισαγγελέα τώρα που είναι στο Βελιγράδι ε, και ποια είναι η αίσθηση για την αξιολόγηση που αυτός θα έχει. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια πρόταση στον πρόεδρο Αλμπερτίνη. Ε, ίσως θα μπορούσε η Επιτροπή να απευθύνει μια πρόσκληση στον κύριο Μπράμερτς να ακούσουμε από πρώτο χέρι την αξιολόγησή του για τη συνεργασία της Σερβίας και να μπορέσει να γίνει πια επί του συγκεκριμένου και να φύγουμε από ε, ιδεολογήματα και κατασκευές οι οποίες έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Νομίζω, Πρόεδρε, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κοπά. Σίγουρα η πρότασή σας θα εξεταστεί. Πιστεύω με ευνοϊκό πνεύμα. Θα το εξετάσουμε. Βάγκελ, για 1,5 λεπτό, κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. 1,5 λεπτό είναι κάπως λίγο για να μπορεί κανείς να παρέμβει σοβαρά. Σας καλωσορίζω ως εκπρόσωπο της νέας γενιάς των Σέρβων πολιτικών. Είμαι πεπισμένος ότι και εσείς, αλλά και ο προκάτοχός σας Φιλάνοβιτς που το είχε ήδη δηλώσει, ότι θα είστε σε θέση να προωθήσετε μια σύγχρονη, μια μοντέρνα Σερβία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που οι νεαροί Σέρβοι θα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη σύντομα, όπως μπορούσαν να το πράξουν και οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους. Χαίρομαι που φαίνεται αυτά να δίνουν και μια θετική κατεύθυνση στην ε, ε, σερβική κοινή γνώμη ε, υπέρ μιας ευρωπαϊκής πορείας. Μιλήσαμε πολύ για το Κόσοβο σήμερα. Μιλάμε βέβαια όμως τώρα για μια χώρα η οποία έχει αναγνωριστεί από 24 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέσω τώρα το θέμα της επιστροφής των Σέρβων στην Κροατία που τα συζητήσαμε και προηγουμένως. Ρωτώ τώρα και συγκεκριμένα σχετικά με την προστασία των Σέρβων στο Κόσοβο και την προστασία των σερβικών μοναστηριών στο Κόσοβο που είναι σημαντικά θέματα και μέσα στη συζήτηση για το Κόσοβο. Εκτιμώ ιδιαίτερα την επίσκεψη Χθε του ε, Προέδρου σας στην Σρεμπρένιτσα. Τονίζω ότι ωστόσο ότι είναι απαραίτητο πια ο Μλάντιτς να αχθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις σας στην αρχή Αναφερθήκατε σε προτεραιότητες της χώρας σας. Πολύ εύγλωτα, όπως είπαν όλοι. Και χάρηκα, διότι θέσατε σωστά τις προτεραιότητες. Πρώτα αναφερθήκατε στο πολιτικό μέλλον της χώρας σας, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βεβαίως, όλοι τώρα περιμένουμε συγκεκριμένες αποδείξεις, πράξεις, ότι πράγματι προχωράτε προς τα εκεί αναφερθήκατε και σε ανησυχίες για ενδεχόμενο διάλειμμα, διακοπή, αφού προσχωρήσει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μία διακοπή των διευρύνσεων λόγω κοπόσεως κλπ. Ο κύριος Κάτσι νομίζω ότι ανέφερε ακροθυγός και θέλω να το επιβεβαιώσω. Μην ενθουσιάζεστε, μην ανησυχείτε όταν ακούτε ομιλίες για αυτή τη διακοπή. Ε, να επικεντρωθείτε στο να εκπληρώσετε, να πετύχετε τα κριτήρια που αφορούν το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας. Αν τα καταφέρετε, κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Όλοι θα πρέπει να το αναγνωρίσουν στο μέλλον. Πολλοί προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στο θέμα που θέλω να θέσω κι εγώ. Ερώτημα, χωρίς επικριτικό πνεύμα, η σερβική κυβέρνηση τι κάνει για να λύσει το πρόβλημα που αποκαλείται Ράτκο Μλάντιτς. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν κυρία Γκόμες, για 1,5 λεπτό. Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζω και εγώ την ομιλία σας και τις ε, εξελίξεις για τις θεωρήσεις. Το ερώτημα τώρα αφορά τις τοπικές εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο. Κανείς δεν περίμενε να συμφωνήσετε να πείτε στους Σέρβους που ζουν εκεί να ψηφίσουν διότι Διαφορετικά θα κρατώνται όμοιροι και δεν θα μπορούν να κάνουν σωστά τη ζωή τους εκεί και να συνεισφέρουν και στη δημοκρατική διακυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου. Όπως είπατε, ξέρετε πόσο επίσης είναι σημαντικό το θέμα του Μλάδη και του Τάτζικ. Εάν όμως οι εγκληματίες πολέμου θέλετε να προσαχθούν στην δικαιοσύνη, γιατί δεν επιτρέψει στη Γιούλεξ να αναπτυχθεί στην περιοχή της Μητροβίτσα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ούτε την ε, ε, Σερβία, ούτε το Κωσυφοπέδιο, ούτε την δικαιοσύνη υπηρετεί. Επίσης, σε θέματα η οικονομία έχετε προβλήματα τύπου που δεν βοηθούν κανένα να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάκη, έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, δεν θα ξαναμπώ σε όλες τις λεπτομέρειες που έφτιαξαν άλλοι συνάδελφοι. Θα απορρίψω ωστόσο ένα πράγμα και μάλιστα αυστηρά που είπατε προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν οι Σέρβοι που η πατρίδα τους είναι το Κόσοβο, που ζουν στο Κόσοβο, που θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές, δεν μπορούν να συγκρίνονται με τους Αλβανούς που βοήθησαν τον Μιλόσεβιτς να πράξει όσα έπραξε. Σας παρακαλώ πραγματικά να τα ανακαλέσετε. Χθε ήρθαν και επισκέφθηκαν 8 νεαροί Σέρβοι στο γραφείο μου με συνοδεία διεθνών αλλοδαπών δηλαδή συνοδών και μου είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές στα ε, νέα αποκεντρωμένα όργανα, στις νέες αποκεντρωμένες κοινότητες και θέλουν να βοηθήσουν να οργανωθεί καλύτερα η ζωή. Απορρίπτω λοιπόν απολύτως αυτήν την σύγκριση με ε, τους Αλβανούς εκείνους οι οποίοι βοήθησαν τον Μιλόσεβιτ να πράξει όσα έφραξε. Σας ευχαριστώ κυρία Πακ για ένα λεπτό Βαζέσκου. Για ένα λεπτό, κύριε Βαζέσκο. Θα είμαι σύντομη, το υπόσχομαι. Κύριε Υπουργέ, πώς υποστηρίζετε τους Ρουμάνους της περιοχής Τιμόκ και τι θα πράξετε για να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Σέρβοι δεν αναγνωρίζουν αυτήν την μειονότητα που είναι περίπου 250.000 ενώ αναγνωρίζουν μόνο τη μειονότητα στο Μπανάτ. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκο. Για ένα λεπτό, Λούνα Τσεκ, για δεύτερη παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, παρόλη μου την υποστήριξη για την ένταξη της ε, Σερβίας στην Ένωση και όλη την αναγνώριση των προσπαθειών σας, Θέλω να καταστήσω ένα πράγμα σαφές. Εγώ είμαι η συγγήτρια ε, του Κοινοβουλίου για το Κόσοβο, όχι για τη Σέρβια, για τη Σέρβια που είναι ο κ. Κατσίν. Και στις ε, προσπάθειε που είχα κάνει παλαιότερα ως ε, αυστριακή βουλευτή, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη που τα πράγματα πήγαν όπω πήγαν με το Κόσοβο και δεν είναι ξεκάθαρα. Αλλά η κατάσταση είναι όπω είναι και συμφωνώ με την κυρία Πακ και εγώ δέχθηκα αυτού του νεαρού Σέρβου Κοσοβάρους και εντυπωσιάστηκα από τι δραστηριότητε που αναλαμβάνουν. Όταν λέτε ότι δεν, είστε, δεν χαίρεστε που δεν μπορείτε να ε, ε, ενισχύσετε τις ε, τοπικές εκλογές και λέτε ότι δεν είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατά τα πράγματα εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Οι ε, τοπικέ εκλογέ στο Κόσοβο σημαίνουν ότι οι Σέρβοι Κωσοβάροι θα μπορούσαν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια του. Είναι δυνατόν λοιπόν για εσά. Και σα ζητώ πραγματικά, δεν ανάγκη να τι υποστηρίξετε ανοιχτά, αλλά ζητήστε από του Σέρβου Κοσοβάρου να συμμετάσχουν, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια του. Όπω θέλετε άλλωστε και οι ίδιοι οι Σέρβοι πολίτε μέσα στη Σερβία να αναλαμβάνουν ευθύνε στο τοπικό επίπεδο. ευχαριστώ. Το, κυρία Λούνατζε και έληξε η συζήτηση. Το λόγο έχετε εσεί κύριε Υπουργέ για να δώσετε τις τελικές ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας το ερώτημα που δεν απάντησα στον προηγούμενο γύρο που αφορούσε το συνοριακό, το μεθοριακό θέμα με την Κροατία. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος. Αργή, ξεκινήσαμε να το συζητάμε. Ποτέ δεν το συζητήσαμε πριν. Το ότι ξεκίνησε η συζήτηση δείχνει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Ε, ε, πιο δύσκολο είναι να ξεκινάει κανείς από το μηδέν, να δούμε πώς θα πάει στο μέλλον. Είναι ενδεχομένως περιπλοκότατο ζήτημα και ελπίζω πραγματικά να επιληθεί και να μην αποτελεί βάρο όσον αφορά άλλε προτεραιότητε, Στο τέλος όλοι θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε τα θέματα των συνόρων θα αποκτήσουν διαφορετική σημασία. Τούτου λεχθέντος και έχοντας συζητήσει πρόσφατα το θέμα των συνόρων, δεν είναι πάντα τέλεια τα πράγματα και στην πράξη δεν είναι όπως είναι θεωρητικά και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες διμερός με την Κροατία τόσο ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο σε τίποτα. Τώρα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις με την Κροατία και απαντώντας στο ερώτημα των προσφύγων σχετικά με τους πρόσφυγες από την Κροατία που τώρα ζουν στη Σερβία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, εξακολουθεί να είναι. Δεν έχει γίνει αρκετή πρόοδος εκεί. Ε, ελπίζουμε στο μέλλον να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Θα γίνει μια μεγάλη διάσκεψη για τους πρόσφυγες τον Φεβρουάριο στο Βελιγράδι. Θα διοργανωθεί μαζί με την ύπατη αρμοστία το ΙΕ για τους πρόσφυγες και ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τώρα ε, ελπίζουμε ότι έχουμε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζουμε να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε συζήτηση στην Κροατία το πρωί. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω συζητώντα την ε, Κροατία. Το δικαίωμα τη επιστροφή των Σέρβων που απελάθησαν από την Κροατία κατά τη διάρκεια της, ε, των επιχειρήσεων των 1995 τη επιχείρηση Storm, όταν εν μία ανοιχτή 250.000 Σέρβοι ε, καθαρίστηκαν από την Κροατία. Η επιστροφή στις πατρίδες τους από όπου εκδιώχθηκαν ε, δεν επιλύθη ικανοποιητικά. Παραδεχόμαστε τις προσπάθειες της κυβερνήσεως της Κροατίας, προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα και θέλουμε να συνεχιστεί συνεργασία μαζί τους και με οποιονδήποτε άλλον, ούτως ώστε Όποιος έχει διωχθεί από το σπίτι του λόγω του χάους της δεκαετίας του 90 να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει πολίτης της Ευρώπης με πλήρη δικαιώματα εκεί που γεννήθηκε. Θα εξακολουθήσουμε τη συνεργασία και με την Κροατία και με όλους τους άλλους πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλοί ρωτούν για τον Μλάντιτς και για αυτούς που, για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου. Προσπαθώ να σκεφτώ τι λησμόνησα να πω στα προηγούμενα σχόλιά μου. Προσπάθησα σκληρά. Αλλά ίσως χρειάζεται και άλλη διευκρίνηση να επαναλάβω κάτι. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε, τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε δεν έχει μείνει, όλα τα κάνουμε. Η ερώτηση ήταν τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τι δεν είναι στα, στις δυνάμεις που έχουμε στα χέρια μας, στις δυνατότητές μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ απάντηση. Ψάχνουμε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται, η οποία γίνεται σε διεθνές επίπεδο αυτή η προσπάθεια. Αν κάποιος έχει κάποια πρόταση, έχουμε τρόπους να εστερνιστούμε την πρόταση και να την εντάξουμε αυτή την πρόταση στην προσπάθεια που καταβάλουμε. Εάν ξέραμε πού είναι, ήταν ο Μλάντιτς, ο Μλάντιτς δεν θα ήταν ελεύθερος. Σας διαβεβαιώνω και σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η θέση μας θα είναι αμετάβλητη μέχρι ότου δεν υπάρχουν ε, κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Καμιά φορά δεν είναι εύκολο να βρει κανείς έναν ο οποίος ήταν ε, αξιωματικός ε, επικεφαλής στρατιωτικών δυνάμεων και είναι κάπου στην Ήπεθρο που κρύβεται. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε τον Μλάντιτς. Τελευταία φορά που τον είδαν, τα τελευταία του ίχνη ήταν κάπου στην Ήπεθρο. Πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και κανεί δεν αμφισβητεί τι προσπάθειες που καταβάλουν. Δεν τον βρήκαν όμω ακόμα. Προσπαθούμε να βρούμε αυτούς τους κατηγορούμενου και δεν θα παραιτηθούμε από αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι είναι σωστό όλοι να περάσουν από δίκη και δεν θα παραιτηθούμε. Τώρα, όσον αφορά την Βοσνία ριζεγοβινη με κάθε σεβασμό να απορρίψω τις κατηγορίες ότι η πρεσβεία της Σερβίας, η πάλι της πρεσβείας της Σερβίας ε, εργαζόταν, κινήθησαν κατά της απελευθέρωσης, της εξαίρεσης θεωρήσεων για τη Βοσνία Ζεγοβίνη που δεν είναι. Αν θέλετε την επίσημη θέση της κυβερνήσεως της Σερβίας πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς απελευθέρωση από τις θεωρήσεις αύριο. Διάλογος εκτός μικροφώνου, δεν ακούνε διερμηνείς, απάντηση του Υπουργού. Θα πρέπει να ακούσετε ποια είναι η επίσημη θέση της κυβερνήσεως, ότι ελπίζουμε πράγματι ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, να έχει το ίδιο δικαίωμα. Οι πολίτες της Βοσνίας Ζεγοβίνης να έχουν το ίδιο δικαίωμα όπως οι πολίτες της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής. Ταχύτερο και αυτό θα ήταν παρακινδυνευμένο να μείνει κανείς εκτός και πίσω. Και αν είχε κανείς ένα μαγικό ραβδί, να το κάνει να συμβεί αύριο για τους πολίτες της Βοσνίας Ρεγοβίνης, κάντε το. Σας συμβουλεύω να το κάνετε. Ανεξάρτητα από προδιαγραφές και όρια. Ξέρω ότι είναι ανέφικτο. Γι' αυτό εγώ μιλούσα για μαγικό ραβδί. Αλλά υπάρχει πολιτική βούληση και είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τα πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσουμε να φτάσουν εκεί το ταχύτερο δυνατόν αντιπαθούμε αυτή την κατάσταση να μην είναι στην ίδια θέση που θα είμαστε εμείς αν θέλει ο Θεός από την 1η Ιανουαρίου. Όσον αφορά τη Βοσνία Ζεγοβίνη, η πολιτική της Σερβίας είναι εξή. Θέλουμε αυτή η χώρα να μείνει ενωμένη, να, να ζει σε ευμάρεια, να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μείνει πίσω αυτή η χώρα. Επουδενή, επουδενή τρόπο να μείνει πίσω. Αυτή είναι η θέση της Σερβίας και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο αυτή η κυβέρνηση έχει την εξουσία. Και όσον αφορά τη Σρεμπένιτσα, να το πω ξανά. Είχαμε τη στιγμή μας Βίλι Μπραντ, τη δέκατη επέτειο του φρικτού, δέκατη επέτειο της φρικτής αυτής, του φρικτού αυτού γεγονότος. Ήταν ο πρόεδρος μας εκεί και ήμουν και εγώ μαζί του και υποκλήθηκε στα θύματα και είπε ξεκάθαρα σαν δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Σερβίας είπε τι σκέφτεται για το θέμα εξελέγει από το λαό, υποστηρίχθηκε από το λαό να ακολουθήσει ένα όραμα και ένα κομμάτι του οράματος ήταν αυτό που έκανε και αυτό που είπε και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που έκανε Ποτέ, ποτέ, σε καμία περίσταση, υπό οποιαδήποτε μορφή δεν μπορούμε να αρνηθούμε, να μειώσουμε, να ξεχάσουμε, να επιτρέψουμε να λησμονηθεί αυτό που συνέβη στη Σρεμπνέτζιτα. Φρικαλαιότητα που αξίζει κάθε καταδίκη. Και ελπίζω σύντομα να βρεθούμε στην κατάσταση με την πάροδο του χρόνου όπου πράγματι θα τα αφήσουμε αυτό πίσω όπως πολλά εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί σε αυτή την Ήπειρο και τώρα έχουν μείνει στο παρελθόν. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Αλλά δεν θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τις ευθύνε μας σχετικά με το θέμα και γι' αυτό θα κάνουμε τη δουλειά όσον αφορά τη συνεργασία με την Χάγη. Λυπούμε που δεν μπορώ να σας δώσω καλύτερη, πιο πλήρη ε, απάντηση ή που δεν μπορώ να σας δώσω τη διεύθυνση, τη διεύθυνση των ε, καταζητουμένων. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα αναπαυθούμε μέχρι ότου αυτό να τελειώσει. Μιλώντας τώρα για τη συνεργασία με την ULEX, να υπογραμμίσω ότι υποστηρίζουμε αυτή τη συνεργασία. Είμαστε δεσμευμένοι να την ακολουθήσουμε τη συνεργασία. Νομίζω ότι η Σερβία αποδεικνύει ότι είναι ίσως ο πιο βάσιμος αξιόπιστος εταίρος από όλου στην Γιούλεξ. Τα οχήματα της Γιούλεξ, η διοκτησία της Γιούλεξ δεν καίγονται, δεν αποτελούν αντικείμενο κλοπής από τους Σέρβους, δεν τα κλέβουν, δεν μάλλον δεν τα πετροβολούν. Οι Αλβανοί τα πετροβολούν και τα κλέβουν. Και τα καίνε. Έγινε και στην Μητροβίτσα και έγινε και στην Πρίστινα και συμβαίνει. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να τα δούμε όλα με προπτική. Η κατάσταση στο κοσυφοπέδιο βελτιώνεται παρά σοβαρές βαθιές διαφωνίες που υφίστανται και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν εν μία νυχτή θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πράγματι η κατάσταση στο κοσυφοπέδιο είναι δύσκολη. Όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, ίσως είναι μία από τις πρωτεύουσε του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Είναι πολύ ατυχής η κατάσταση, αλλά η Σερβία δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτό το οργανωμένο έγκλημα εκτός από συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με το ψήφισμα 244 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και συμφωνώ μεν ότι η κατάσταση στη Μητροβίτσα πόρα έχει από το ιδεώδες. Επίσης όμως θα ήθελα να πω ότι άλλα μέρη του κοσυφοπεδίου, ε, σε άλλα μέρη ίσως είναι να είναι χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά λαθρεμπόριο, οργανωμένο έγκλημα, πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν και όλοι θα πρέπει και ελπίζω και εύχομαι να προσπαθήσουν όλοι να εξαλείψουν από προσώπου, από προσώπου της επαρχίας αυτά τα προβλήματα. Η κατάσταση όσον αφορά την ε, ιδιοκτησία της εκκλησίας, εκκλησιαστική διοκτησία και τις ε, σερβικές ε, εκκλησίες στο Κωσυφοπαίδιο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Θέλω να πω ότι κινδυνεύουν μοναστήρια από το Μεσαίωνα, παγκόσμια κληρονομιά, που αντιμετωπίζουν ε, πολύ δύσκολη κατάσταση και κινδυνεύουν τα μοναστήρια. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο Κωσυφοπαίδιο. Ίσως να Ακούσατε για το μοναστήρι Ντέτσεν, ένα από τα παλιότερα, τα ομορφότερα μοναστήρια, μεσαιωνικά σερβικά μοναστήρια, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO που κινδυνεύει. Υπάρχει επανειλημμένη άρνηση να επιστραφούν τα περιουσιακά στοιχεία ε, του ε, μοναστηριού. Ακόμα και όταν η διεθνής κοινότητα έδωσε εντολή στην αλβανική, στις αλβανικές αρχές να το κάνουν, ε, δεν έγινε και εξακολουθεί η κατάσταση να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ήθελα να θέσω κάτι που έθεσα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας επανειλημμένα. Υπάρχει Τσακοβίτσα. Στο κέντρο της πόλης υπήρχε μια εκκλησία. Δεν υπάρχει πια. Ξέρετε τι έγινε. Την κάψανε. Και τη στρώσαν από πάνω και την κάνανε πάρκο. Στο κέντρο της Τσακοβίτσα, εκεί που ήταν η εκκλησία. Λοιπόν, η εξαφάνιση κάθε ίχνους ύπαρξης της Εκκλησίας. Αυτό έγινε. Το έθεσα τρεις φορές στο Συμβούλιο Ασφαλείας το θέμα. Το θέσαμε στην UNESCO και το θέτω και εδώ το θέμα. Αυτό είναι ο δρόμος για τη συμφιλίωση. Να καίνε και να καταστρέφουν εκκλησίες και μετά να τις στρώνουν από πάνω, ασφαλτοστρώνουν, να κάνουν πλατείες, να κάνουν δημόσια πάρκα από πάνω. Δεν νομίζω ότι αυτή, αυτός είναι ο δρόμος. Συγγνώμη που απαντώ συναισθηματικά σε αυτό το ερώτημα, αλλά ακριβώ έτσι αισθάνεται ο σερβικός λαός για τις εκκλησίες στο Κωσυφοπαίδιο. Πολλοί από εσά ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερα ε, ε, ιστορικά και θρησκευτικά συναισθήματα απέναντι στο Κωσυφοπαίδιο και υπήρξαν και άλλες δύο ερωτήσεις που αφορούσαν τη ρουμανική μειονότητα. Συνεργαζόμαστε στενά με τη ρουμανική μειονότητα. Είναι ένα, ένα κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι στενή εταίρη. Υπάρχει καλή στενή συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ Σέρβων και Ρουμάνων, όχι μόνο στη Σερβία αλλά και στη Ρουμανία και οπουδήποτε στον κόσμο. θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία ούτω ώστε καμία εθνοτική μειονότης και είναι και η ρουμανική μειονότητα ανάμεσα σε αυτές να μείνει σε δύσκολη θέση στη Σερβία. Καμία μειονότητα. Όσον αφορά την προστασία των εθνοτικών μειονοτήτων, η Σερβία μπορεί να ισχυρίζεται ότι η νέα Σερβία, ότι ηγείται, η δημοκρατική Σερβία που εκπροσωπώ, κοιτάξτε τι γίνεται στη Βοηβοδίνα, είναι σαν μια Ευρώπη σε σμίκριν